Φίλοι, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εγώ τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος Μπούζεκ θα έρθει εντός ολίγου και του υποσχέθηκα να ξεκινήσω εγώ τη συνεδρίαση και να αρχίσουμε να συζητάμε τα θέματά μας. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης την έχετε στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς αλλαγές. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει κάτι, επομένως εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ε, ακυρώσουν την συνεδρίαση της Δευτέρας 13 ε, Απριλίου από τις 3 έως τις 6.30 αλλά η συνεδρίαση της Τρίτης της 14ης Απριλίου θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί. Η δημόσια ακρόαση για την εσωτερική αγορά ενέργειας για την Ενεργειακή Άνωση η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 13 Απριλίου θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου σε μια νέα ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις μας. Η σημείο υπαριθμών 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 3ης ε, και 4ης Δεκεμβρίου του 2014 και αυτά τα πρακτικά τα έχετε στους φακέλους σας και αν δεν υπάρχουν σχόλια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά, επομένως εφόσον δεν βλέπω σχόλια εγκρίνονται. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρήπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθου μονάδε καύση. Όπω γνωρίζετε, η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι ένα διαμεθοριακό πρόβλημα και πολλά κράτη-μέλη ε, εισάγουν σημαντικό τμήμα των ε, ρηπών του από τι γειτονικέ χώρε και επομένω χρειάζεται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνεπέ φιλόδοξο πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τι εκπομπέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ε, πληρώσει ένα πολύ σημαντικό κενό ε, για τα μικρά ε, μονάδες τάσης και τις μεγάλες μονάδες τάσης, οι οποίες αυτή τη στιγμή ρυθμίζονται μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες τάσης. Έχουμε προβλέψει μισή ώρα συζήτηση για το θέμα αυτό και να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φέντερλε. Παρακαλώ. το, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την ανάλυση των καθηκόντων σας, έστω και προσωρινά. Ε, νομίζω ότι έχετε λάβει όλοι το ε, κείμενο της νομοδότησης. Ε, θα σας πω δύο λόγια του περιεχομένου. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, όσον αφορά τους ρήπους και την ατμοσφαιρική ρήπανση, πολλές χώρες μας εισάγουν τους ρήπους τους ε, από τις γειτονικές χώρες. Προσπαθώ να βρω μια ισορροπία μεταξύ αυτών των οποίων προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των όσων δήλωσε και το Συμβούλιο μετά τη συνεδρίασή του. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο. Η σχέση με την κείμενη νομοθεσία, επί παραδείγματι, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει διπλή ρύθμιση για τις μονάδες καύση. Υπάρχει ήδη νομοθεσία ενισχύ για τις μεγάλες μονάδες καύση. Ε, δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ε, ε, έχουν τις μικρές μονάδες καύση. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού. Το δεύτερο στοιχείο είναι να μην υπάρχει υπερβολική νομοθεσία, διότι ε, όπως είπα κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ασχολούνται με τις ε, μεσαίου μεγέθους και τις μικρού μεγέθους μονάδες καύσης. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κόστους για τις επιχειρήσεις και τα ε, στοιχεία και την υγεία και τι ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το δούμε και αυτό και μέσω τροπολογιών. Επίσης εξετάζουμε και το θέμα της ευελιξίας για τις μικρότερες μονάδες. Ε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τις μικρότερες μονάδες ότι μπορεί να υπάρχει υπερβολική νομοθεσία και θέλουμε να έχουμε λίγη μεγαλύτερη ευελιξία από όσοι παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασχολήθηκα επίσης και με κάποιες από τις εξαιρέσεις που παρουσίασε το Συμβούλιο. Ήταν αρκετές αυτές και ε, θεωρώ ότι πρέπει να περιοριστούν. Νομίζω ότι θα υπάρξουν αρκετές τροπολογίες από του σημείου αυτού, αλλά είμαι διατεθειμένος φυσικά να το συζητήσω το ζήτημα, διότι με καλά επιχειρήματα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Προσπαθώ να τονίσω και με κάποια λεπτομέρεια, διότι είναι και πολύ τεχνικό το ζήτημα ε, για τα διάφορα επίπεδα εκπομπών και υπάρχουν διάφορες απόψεις επί του σημείου αυτού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, κατάλληλο πλαίσιο, να μην υπάρχει υπερβολική νομοθεσία, να μην υπάρχει διπλή ρύθμιση για τις μονάδες καύσης και επίσης να ε, αντιληφθούμε και ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα παραγωγικό τομέα ε, ο οποίος θα συνδυάζεται και με την ενεργειακή ασφάλεια, ε, διότι διαπιστώνουμε ότι σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στις χώρες της Βαλτικής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και ε, το συνδυασμό με τα ωφέλη για το περιβάλλον, παραδείγματο χάρη βιοκαύσιμα για αυτές τις μονάδες καύσης. Ε, αυτά λοιπόν και θα ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις των σχεδόν συγητών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φέτερλε να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στους πιο δυσηγητές. Ο κύριος Ρόιλ από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Φίντερλάι. Ε, ήδη μπορέσαμε να τα πούμε μεταξύ μας και θέλω να σας πω τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχαμε πολύ καλή συνεργασία, όπως βέβαια και με τους άλλους και ηγητές. Και αυτό είναι απαραίτητο διότι η πρόταση της Κομισιόν και κατά τη δική μου άποψη παρουσιάζει προβλήματα. Ε, ελοχεύει ο κίνδυνος ε, της ε, επικάλυψης των ρυθμίσεων ή άλλων περιττών κανονισμών. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν θέλει κανείς να επιτύχει κάτι καλό, τι είναι να υπερβάλλει. Και αυτό όμως είναι σε αντίφαση με αυτά που προτίθεται να κάνει η νέα επιτροπή, η οποία θέλει να προσέχει πάρα πολύ το τι ακριβώς θα ρυθμίζεται. Σπάνια έχει υπάρξει τέτοια πρόταση που να δέχεται τόσο έντονη κριτική και αυτό φαίνεται επίσης από το ότι στο Συμβούλιο που συζητεί το θέμα και το είπε ο κύριος Φέντελε, στο Συμβούλιο λοιπόν έχει κατατεθεί μια μεγάλη σειρά τροπολογιών οι οποίες πρέπει να πω είναι πάρα πολύ καλές. Η προσέγγιση του Συμβουλίου, κατά την άποψή μου, είναι πολύ πιο έξυπνη από αυτήν της Κομισιόν και αυτή είναι μια πρόταση που σπάνια τη βγάζω από το στόμα μου, αλλά στην περίπτωση ισχύει. Μία λοιπόν από τις προτάσεις ε, του κειμένου του Συμβουλίου την έχει ήδη υιοθετήσει ο εισηγητής, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε και το βρίσκω πολύ θετικό ε, το ότι τόσο ο Συμβουλίο όσο και η Κομισιόν ε, λαμβάνει υπόψη της ε, τα ανώτατα και τα κατώτατα αέρια των ε, μονάδων αυτών ε, κάψεως ή το ότι διευκολύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Για μένα υπάρχει ένας κίνδυνος, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος επικάλυψης ρυθμίσεων, γι' αυτό και λοιπόν θα καταθέσω μια πρόταση για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς. Και θέλω να πω και το εξή. Βεβαίω δεν αρκεί να πει κανείς στην Κομισιόν τα πιο ε, σαφή γιατί εμείς πρέπει να το πράξουμε αυτό. Εμείς πρέπει να ορίσουμε σαφή Η οδηγία MCP ισχύει για εγκαταστάσεις 1 μέχρι 50 ΜΒ. Από 50 ΜΒ ισχύει η οδηγία περί εκπομπών της βιομηχανίας που υπάρχει. Ε, αν λοιπόν θέλουμε να ρυθμίσουμε κάτι, τότε να μην ρυθμίσουμε αυτό που έχει ήδη ρυθμιστεί. Και κάτι άλλο. Στην πρόταση Κομισιόν γίνεται λόγος ε, για σκόνη, λεπτή σκόνη αυτό αναμφίβολα θα δημιουργήσει νομική ασάφεια. Το Συμβούλιο λοιπόν αυτή τη λεπτή σκόνη την μετονομάζει σε σκόνη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δεχτούμε ως Κοινοβούλιο. Η άλλη πρόταση που κατά την άποψή μου είναι ενδιαφέρουσα είναι η εξή. Το Συμβούλιο ορίζει λογικές εξαιρέσεις όπως για υπερπόνητες περιοχές και άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν προβλήματα ατμόσφαιρας. Εξάλλου υπάρχει και η υποχρέωση δήλωσης για τα κράτη-μέλη, η υποχρέωση η δέσμευση για, κράτη για μονάδες οι οποίες πρόκειται να κλείσουν και μια ρύθμιση της Κομισιόν για ειδικέ περιοχές όπου ξεπερνιόνται τα ανώτατα όρια που ισχύουν για την ατμόσφαιρα. Αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Πάντως μπορώ να καταλήξω και επανέρχομαι στην αρχική μου παρατήρηση ότι η πρόταση Κομισιόν είναι προβληματική, το Συμβούλιο κατέθεσε προτάσεις που κατά την άποψή μου μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση και θεωρώ επίσης ότι πολλές από τις κατατεθήσεις προτάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Οι περισσότερες εξ αυτών ε, είναι του εισηγητή. Εγώ αργότερα θα καταθέσω συγκεκριμένε τροπολογίες και στην ψηφοφορία θα μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε περιττέρω. Θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερα αν η Κομισιόν είχε κάνει τη δουλειά της με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρόιλ. Η κυρία Κούμπα Νάτρη από τους σοσιαλδημοκράτες. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Εύχομαι σε όλους σας ε, καλή εβδομάδα μετά τις ε, διακοπές. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φέντερλε. Πήραμε το έγγραφό του έγκαιρα, του ρίξαμε μια ματιά και μπορούμε πάνω σε αυτό να δουλέψουμε. Ε, και εγώ ε, πήρα περίπου τα ίδια μηνύματα όπως και ο προλαλής σας. Έτσι λοιπόν, εφόσον μιλάμε για την δυνατότητα να μιλάμε για βιοενέργεια, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εφόσον μιλάμε και για την καθαρότητα του αέρα, είναι δύσκολο να βάλει κανείς το σύνολο της Ευρώπης μέσα σε ένα καλούπι, γιατί υπάρχουν και πολύ διαφορετικές περιοχές υπάρχει οδηγία περί ε, περιορισμού των εκπομπών. Αυτή κατατέθηκε πολύ έγκαιρα και θα ολοκληρωθεί και πολύ νωρίτερα. Διότι οι εκπομπές των μικρομεσαίων μονάδων καύσης ε, στην Ευρώπη είναι κάτω από το 5% όλων των εκπομπών και έτσι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Βεβαίως ελπίζουμε στην Ευρώπη η ποιότητα του, της ατμόσφαιρας να είναι καλύτερη, καθαρότερη και να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις εκπομπές. Να σας πω λοιπόν, ε, μάλλον στις λεπτομέρειες, θα μπω τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Νομίζω ότι το δικό μας ε, το καθήκον στην Επιτροπή είναι ακριβώς να προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους μας. Έχει μείνει ακόμα αρκετή δουλειά ε, σχετικά με τους ε, και πώς μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλό κονισμό. Ο κ. Φέντερλε έχει ήδη κάνει προτάσεις σχετικά με τη χρήση, την καλύτερη χρήση της βιοενέργειας και το Συμβούλιο μετά την Επιτροπή διευκρίνησε ορισμένα θέματα. Εγώ είμαι πολιτικός από τη Φινλανδία. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, συγκεκριμένε διατάξει για τα δάση στη δική μα την περιοχή. Είναι λοιπόν δύσκολο να μιλάμε εδώ ε, για το πώ μπορούμε να χρησιμοποιούμε ενέργεια και κυρίω πολύ δύσκολο είναι το θέμα τη βιοενέργεια. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή οδηγία ε, που θα την διαβάσουμε περαιτέρω γιατί δεν είμαστε η τελευταία επιτροπή που γνωμοδοτεί. κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ο κύριος Γκομπάτσεκ ε, από τους ε, συντηρητικού συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί μας παρουσίασε μια πολύ καλά προετοιμασμένη έκθεση. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω μία λεπτομέρεια, κυρίως αναφορά αυτές τις ε, μικρές αλλά και τις ε, μικρομεσαίες ε, μονάδες, εκεί για τις οποίες δεν υφίστανται ακόμα κανονισμοί. Οι κανονισμοί λοιπόν οι οποίοι αφορούν αυτές τις, αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, αυτοί οι κανονισμοί προσφέρουν πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τη γεωθερμία και με αυτόν τον τρόπο να ε, λειτουργούμε τις μονάδες. Ε, ο κύριος Φέντερλε αναφέρει ότι αυτό μπορεί να είναι ε, κίνδυνος, ε, αλλά επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει ε, να εξευρεθούν ειδικέ λύσεις για αυτές τις μονάδες που χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα κάψιμα, βεβαίως μονάδες κάψης μέχρι 5 ΜΒ το μεγαλύτερο κομμάτι της έκθεσης το στηρίζουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε απόλυτα, κατά 100%. Βεβαίως αυτό που έχει επίσης σημασία είναι από κοινού να αναζητήσουμε λύσεις ε, στην Επιτροπή μας με την εξής έννοια, ότι αυτά τα οποία θα πούμε να υποστηριχθούν και από το υπόλοιπο Κοινοβούλιο. Ε, αν θέλει και κάποιος άλλος ε, ο μπορεί να ζητήσει το λόγο για σύντομη παρέμβαση. Ε, παρακαλώ. Δεν έχω εγώ. Δεν, έχω. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Κομπατσίκ. γιατί πιστεύω κι εγώ ότι η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει ο εισηγητής είναι πολύ λογική. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δεν προσφέρεται για πειραματισμούς ή εξαιρετικά ε, γρήγορες και ριζικές αλλαγές που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν και σε προβλήματα. Στην περιοχή από την οποία προέρχομαι είναι ένα ζήτημα το οποίο μας, ε, αφορά γιατί έχουμε δεκάδες ίσως και εκατοντάδες μονάδες τέτοιες μικρής καύσης οι οποίες χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην δημιουργηθεί ανταγωνισμός χωρίς λόγο μεταξύ όμορων κρατών. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον υποστηρίζω πλήρως. Σας ευχαριστούμε κυρία Βίρκολα. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή ε, Βιομηχανία. Επομένω, πρέπει να έχουμε υπόψη μα την οπτική γωνία τη βιομηχανία. Βεβαίω, η ποιότητα τη ατμόσφαιρα και του αέρα είναι πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ποιο είναι το κόστο για τη βιομηχανία να υιοθετήσει αυτέ τι ε, αλλαγέ και άρα χρειάζεται να γίνει μια αξιολόγηση του κόστους και του ωφέλου από τον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρήπων. Γνωρίζω από την εμπειρία της Φιλανδίας ότι το σημαντικό η... ο αριθμό που μα δίνει η Επιτροπή για τι μικρέ μονάδε είναι 400, πιθανώ να είναι πολύ περισσότερε, μπορεί να είναι 4.000. και πιστεύω ότι σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές όπου δημιουργείται πρόβλημα ε, για την, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ίσως θα έπρεπε οι χώρες αυτές να έχουν τη δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο να περιορίσουν τη δημιουργία τέτοιων μονάδων, ίσως εκείνες τις περιοχές να μην είναι και τόσο ε, σκόπιμο να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες. Καλύτερα λοιπόν πέρα από το ευρωπαϊκά όρια να δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη στι περιοχέ εκείνε που υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα να υιοθετήσουν πιο αυστηρά κριτήρια, πιο αυστηρού κανόνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον Τζανονάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε γενικέ γραμμές συμφωνώ με τη γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι είναι καλογραμμένη και λαμβάνει δεόντω υπόψη και το βασικό στοιχείο, δηλαδή το γεγονό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι περί αυτών πρόκειται, κινδυνεύουν με πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό ε, άκθος εάν εφαρμόσουμε για αυτές ε, τα ίδιους κανόνες που εφαρμόζουμε και για τις μεγάλες μονάδες καύσης. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Αυτό όμως που μου προξενεί περιέργεια κάθε φορά που διαβάζω τέτοιες ε, γνωμοδοτήσεις είναι τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται και δεν καταλαβαίνω και από πού προέρχονται. Τι ακριβώς εννοώ. Από πού προκύπτει ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση προκαλεί 400.000 πρόωρους θανάτου ετησίως μου φαίνεται ότι πρόκειται για ένα στοιχείο ότι μάλλον είναι επινόημα από κύμα της φαντασίας μας, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις επ' αυτού και δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ ενός πρόωρου θαλάτου από κάποιον άλλον. Ή το γεγονός ότι δίνονται 40 δις ευρώ για κόστος για την υγεία. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακριβές αυτό το στοιχείο ή δίνουμε έτσι λίγο αφαίρετα στοιχεία. Τέλος, λέει ότι αν η Κίνα δεν είχε ατμοσφαιρική ρήπανση, θα είχε ένα καθάριστο εγχώριο προϊόν ε, κατά 12 με 13 ποσοστίες μονάδες ανώτερο. Δηλαδή θα είχαμε ένα ΑΕΠ στην Κίνα που θα ήταν πάνω από το 25%. Σας παρακαλώ, αυτά τα στοιχεία να τα αναφέρουμε λίγο πιο προσεκτικά, διότι οτιδήποτε μπορεί να έχει συνέπεια για τη ε, ζωή των πολιτών μας θα πρέπει να αναφέρεται με πηγές για να μην έχουμε στοιχεία τα οποία δεν θα έχουν καμία επιστημονική ε, επιβεβαίωση. Έχουμε πάνω πολλέ περιπτώσει στις οποίες αναφέρονται κάποια τυχαία στοιχεία και τα, στη συνέχεια αυτά διαψεύδονται. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. please. One minute. Ο κύριος για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, τον Φρέντερικ, για την γνωμοδότηση. Εγώ θα σημείωσω κάτι που είπαν και άλλοι ότι αυτό που αναφέρεται και στην ε, γνωμοδότηση είναι το στοιχείο δηλαδή του ότι το 75% ε, των μεσαίων μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης τελούν υπό τη διαχείριση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τους ε, επιβληθεί υπερβολικός διοικητικός, διοικητικό άχθος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα των μεγαλύτερων εταιριών να προσαρμόζονται και να εκτελούν στι τις απαραίτητες διαδικασίες. Το δεύτερο σημείο σύντομα ε, είναι γεγονός ότι ε, πέραν από τις μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλο μερίδιο ε, της εκπομπής των ρήμων στην ατμόσφαιρα έχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Η ΕΠΑ και η Κίνα και ιδιαίτερα σε τέτοιες οικονομικές συνθήκε, αυτοί είναι που πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο με μειώσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να στρέψει την προσοχή της και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. And then finally, Mr. Tamburano. Ευχαριστούμε κύριε Σταμποράνο. Γεια σα. Πρόκειται για μια πρόταση οδηγίας η οποία λέει ότι θα πρέπει να μειώσουμε και τους ρήπους των ε, ε μεσαίου μεγέθους ε, εγκαταστάσεων καύσης διότι φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ζουν 8 μήνες λιγότερο λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Πολύ ωραία ιδέα θα φαινόταν, αλλά για μα αυτή η πρόταση οδηγία είναι στην πραγματικότητα απάτη, διότι αφήνει να ξεφεύγουν ρηπογόνοι παράγοντε από όλε τι μεριές και πρόκειται για μία δέσμη μέτρων ε, οδηγιών που πρότεινε η Επιτροπή Μπαρόνροζο, που η Επιτροπή Γιούνκερ έχει προτείνει να αποσυρθούν, αν και δεν είναι σαφέ ακόμα αν θα γίνει αυτό ή όχι. Η πρόταση οδηγία έχει κάποιο μέλο ναι. ή επειδή είναι από τι προηγούμενε πολιτικέ ελοχεύει ο κίνδυνο να βρεθεί στον κάλαθο των αχρήστων. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Το Συμβούλιο πριν από εμά εξέτασε αυτή την πρόταση οδηγία και έχει αποφασίσει επί ποια βάση θα ξεκινήσει για τη διαπραγμάτευση. Από το Συμβούλιο έχει προκύψει ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά αποδυναμώνει συστηματικά ε, τι διάφορε διατάξει οι οποίε έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία τη υγεία των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο να εργαζόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Οτιδήποτε προκύπτει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας έχει αποστείλει σαφές μήνυμα ότι ό,τι και να λέμε δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Ε, το γεγονός ότι έχουν ξαναγράψει ουσιαστικά το κείμενο το οποίο έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει ότι αυτό το κείμενο που συζητούμε εμείς είναι ήδη παροχημένο. Επίσης, όσον αφορά την υγεία των πολιτών, για μας αυτό είναι διαπραγμάτευτο και εμείς, τουλάχιστον η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκω, δεν δέχεται να μην ζούμε με πλήρη υγεία σε αυτή τη σύντομη ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Διάβασα το σχέδιο γνωμοδότησης και θεωρώ ότι ε, ουσιαστικά ε, δεν μπορεί να είναι ισχυρό ενώπιον των θέσεων που εξέφρασε το Συμβούλιο. Θα προτείνουμε τροπολογίες με επικοδομητικό πνεύμα για να βελτιωθούμε, διότι θα πρέπει Διακόπτει ο πρόεδρο. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έχω τρία λεπτά. Οι άλλοι μίλησαν πολύ περισσότερο από μένα. The shadow rapporteurs did. Yes. Λαμβάνοντα Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, θα προτείνω τροπολογίες με επικοδομητικό πνεύμα για να βελτιώσω λίγο και ε, υπό το πρίσμα της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκω. Θα πρέπει να μειώσουμε στα 20 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο την ε, κομπή ε, σκόνης και οι μικρές εγκαταστάσεις καύσης θα πρέπει να διέπονται από το πρωτόκολλο του Γκέτεμπορ που λέει η γνωμοδότηση ότι θέλουμε να θέσουμε ενισχύ. Ενώ στην πραγματικότητα προσφέρει προσφέρει διάφορες διεξόδους. Θα πρέπει να μειώσουμε τι παρεκκλήσει που υπάρχουν στο άρθρο 4 για την καταχώρηση των εγκαταστάσεων και να λάβουμε υπόψη τα χαμηλότερα ε, επίπεδα σε περιοχέ, οι οποίε είναι ιδιαίτερα ε, μολυσμένες. Ε, Επίση, θα πρέπει να γίνεται κατάλληλο έλεγχο σε διάφορε εγκαταστάσει, διότι υπάρχουν τεχνολογίε φίλτρου Διακόπτηκε πάλι ο πρόεδρο. Με διακόψατε, με κάνατε να χάσω 30 δευτερόλεπτα. Δεν σέβεστε το γεγονό ότι είμαι σκιώδη εισηγητή και ε, διαμαρτύρομαι επισήμω για τον τρόπο με τον οποίο προεδρεύεται και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Thank you. And now for the Commission, Mr. Christopher Allen, please. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο κύριος Christopher Allen. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς Επιτροπής Θέλουμε να κάνουμε κάποιες ε, παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν τα μέλη να εξετάσουν καλύτερα αυτήν την πρόταση. Εξετάζοντα λοιπόν αυτή την πρόταση, εμείς εξετάσαμε και μία σειρά εναλλακτικών λύσεων ε, που θα μπορούσαν να αφορούν τις ε, μονάδες καύσης για τις οποίες μιλάμε. Και όσον αφορά το κόστο, εκεί υπάρχουν πολλέ δυνατότητες. Επειδή οι περισσότερες εγκαταστάσεις ε, που χρησιμοποιούν ε, αυτές οι περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις, θεωρούμε ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι να περιοριστεί όσο δυνατόν περισσότερο το διοικητικό κόστος, κυρίως για τις ε, μικρές μονάδες. Η διαφορά συμμόρφωσης ανάμεσα στα, στις υψηλές προδιαγραφές που ισχύουν σε κάποια κρατημέλη και στην πρόταση της Κομισιόν είναι επί 8. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε έναν κανονισμό ισόρροπο, αναλογικό αν θέλετε, ε, κυρίως για τις ε, μικρές ε, μονάδες, στην πρώτη τασή μας, έχουμε περιορίσει έλεγχο για κάθε τρία χρόνια. Ξέρουμε και από το σπίτι μας που χρησιμοποιούμε θέρμανση, ελέγχουμε το σύστημα κάθε χρόνο, αλλά εδώ μια φορά τα τρία χρόνια για τις μικρές μονάδες φτάνει. Όσον αφορά τώρα ε, στην ε, συνεισφορά αυτής της ε, πρότασης, τη μείωση της ρήπανσης από τη στιγμή που αυτές οι μονάδες αντικατοπίζουν το 5% της ρήπανσης, επειδή κατά το παρελθόν δεν είχαν ρυθμιστεί τα θέματα, μπορεί να υπάρξει μεγάλος περιορισμός του κόστους και αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα 20 με 22% προστατιών που θα καταβληθούν στο πλαίσιο της προτινόμενης πολιτικής. Όσον αφορά τώρα σε αυτά τα 400.000 άτομα που πεθαίνουν νωρίτερα από ό,τι θα πέθαναν αν δεν υπήρχε η ρήπανση της, του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό βασίζεται περισσότερο σε επιδημιολογικές μελέτες και όχι στον ΠΟΕ, οι επιδημιολογικές μελέτες τεκμηριώνονται, είναι οι καλύτερες και περιλαμβάνονται και στην αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με τη ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα που υπάρχουν. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Το εξή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στον έλεγχο της ρήπανσης και κινδυνεύει να χάσει αυτή την πρωτοπόρο θέση από τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ασία. Αυτή λοιπόν η οδηγία είναι μία από εκείνες οι οποίες ε, θα βοηθήσουν, θα πείσουν τη βιομηχανία ότι αξίζει τον κόπο να παραμείνουν στη θέση που είναι στη διεθνή αγορά. Δηλαδή να αναπτύσσονται ταχύτατα στο Πεκίνο, ας πούμε, τα επόμενα πέντε χρόνια θα επενδυθούν πέντε δις για τον έλεγχο του ατμοσφαιρικού αέρα, που είναι πολύ περισσότερα από ότι στο σύνολο της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν μιλάμε για μεγάλες αγορές και για μεγάλες μονάδες. Ελπίζω λοιπόν με τα σχόλιά μου να παρουσίασα, να έφτιαξα τα βασικά θέματα, αλλά αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση, παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Φέντερλη, παρακαλώ, για να ολοκληρώσετε το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους τους ισκαιοδησηγητές και τα μέλη της Επιτροπής ε, για τη γνώμη που εκφράσετε. Τα σημείωσα όλα αυτά και θέλω να σας πω ότι είμαι σίγουρος ότι στην Επιτροπή θα επιτύχουμε μεγάλη πλειοψηφία Ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ε, προσβλέπω με χαρά στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Όσον αφορά τα στοιχεία, θα περισπίστηκε λιγάκι η Επιτροπή, αλλά θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία ε, παρουσιάστηκαν και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, είναι του 2011 και θεωρούνται επίσημα στατιστικά δεδομένα της Κομισιόν. Δεν είναι τυχαία τα στοιχεία αυτά και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, γιατί αν κρίνουμε, επικρίνουμε ε, αυτά που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν έχουμε και πολλά πια να πούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά δίνουν έτσι μια ευρύτερη εικόνα από τον που συζητάμε. Αν λοιπόν δεν λάβουμε υπόψη μας το τι ακριβώς, και ε, είναι οι αρνητικές συνέπειες ε, αυτής της μόλις σε εμά, είναι ότι απλά μετακυλίουμε την δαπάνη στο φορολογούμενο που πρέπει να καταφύγουν στο γιατρό και ούτω καθεξής. Ε, Βεβαίω πρέπει να είμαστε σωστοί με του αριθμού, αυτό είναι σωστό. Ε, δεν πρέπει αυτές τις 400.000 θανάτους το 2011 να τις συνδέσουμε άμεσα με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορούν το σύνολο των εκπομπών και από αυτοκίνητα και από άλλους φορείς. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ συνάδελφοι και είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθουμε με μια πολύ καλή ψηφοφορία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ ε, και να σας πω ότι η διορία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 26 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στις 12. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο υπαριθμών 4 και πάμε στο 5 που θέλω να σας πω είναι μεγάλη χαρά για μας το ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο, κύριο Τίμερμανς, ε, για καλύτερους οργανισμούς για το κράτος δικαίου και για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρώτος Αντιπρόεδρος, κύριος Τίμερμανς, ε, θα μας παρουσιάσει το θεματολόγιο για την καλύτερη εφαρμογή κανονισμών, κυρίως ε, κάτω από το πρίσμα των θεμάτων που αφορούν στην Επιτροπή μας. Σας καλωσορίζουμε. Είναι μεγάλη τιμή για μας που ήρθατε. Προσβλέπουμε τις ε, παρατηρήσεις και προβλέπετε επίσης μία ώρα για τη συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως η παρουσίασή μου θα είναι σύντομη. Γιατί ο λόγος που ζήτησα την συνάντηση με την Επιτροπή σας ήταν ε, κυρίως για να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Επομένως θα προσπαθήσω να περιγράψω ε, συνοπτικά τις προτεραιότητες της Επιτροπής αυτή τη χρονιά. Αλλάξαμε τον τρόπο εργασίας ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί διεξοδικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει περιοριστεί για το 2015 λοιπόν το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις δραστηριότητες εκείνες τις οποίες θα υλοποιήσουμε το 2015 και μόνο. Ανακοινώσαμε λοιπόν, μάλλον θα παρουσιάσουμε σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις αποφάσεις μας σε σχέση με τις αποφάσεις που θα αποσύρουμε και φυσικά πιο αναλυτικά το, πρόγραμμα, το λεγόμενο πρόγραμμα Juncker για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Για τα ζητήματα που αφορούν στην Επιτροπή σας, έχουμε ξεκινήσει την εργασία μας για την Ενεργειακή Ένωση, ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένη της ανησυχίας των Ευρωπαίων πολιτών για την εσωτερική ασφάλεια. Ε, προσπαθούμε να, να βελτιώσουμε την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τα κράτη και εκείνα τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας. Θα ήθελα να συγχαρώ να εκφράσω την χαρά μου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε και έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνεχίσει ε, την, την, την, την ε, διαπραγμάτευση για την ανταλλαγή στοιχείων PNR, τα στοιχεία των επιβατών, με αυτόν τον τρόπο δημιουργώντας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες μας στον χώρο Σέγγεν. Και για μένα προσωπικά είναι σημαντική προτεραιότητα η βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να φροντίσει η Ευρώπη να μην μένει πίσω σε σχέση με άλλα κράτη του κόσμου που ε, έχουν βρεθεί πιο μπροστά, έχουν προχωρήσει περισσότερο στα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να σας παρουσιάσει ένα σχέδιο για την κυκλική οικονομία, για την διαχείριση των απορριμμάτων αλλά όχι απλώς τη διαχείριση των απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση ε, υλικών μετά το τέλος ζωής. Και τον τρόπο με τον οποίο θα φροντίσουμε ε, ε, υλικά που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα να μην εισάγονται στο, στο, στον κύκλο. Επίσης, καλωσορίζω την συζήτηση που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε Θέλω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να συνεργαστώ με το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε αυτή τη ε, συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να είναι και πιο αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο καταρτίζουμε την νομοθεσία. Αυτό ισχύει επίση και, και ιδιαίτερα θα έλεγα για τι ε, εφαρμοστικέ πράξει και τι πράξει κατά τη Σα ευχαριστώ. Ε, προσπάθησα να είμαι σύντομο γιατί ήθελα να ακούσω περισσότερα τα δικά σα σχόλια. Ο Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Τίμερμαντ. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Πίμπαλ. Herr herzlichen Dank. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας ε, και θα μιλήσω γερμανικά γιατί καταλαβαίνετε εσείς ε, κύριε Τιμερμάνης πάρα πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θετικά στοιχεία που πρέπει να τα αναφέρουμε αποδίδοντάς σας τα έψημα με την έννοια ότι εσείς ως αντιπρόεδρος θα είσαστε στο μέλλον αρμόδιος για την better regulation, τις, ε, τις καλύτερες ρυθμίσεις, τους κανονισμούς και οποτεδήποτε πρόκειται για θέματα γραφειοκρατίας, η ελπίδα μας είσαστε εσείς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τολμήσατε σε κάποια συγκεκριμένα θέματα να βάλετε και μία διορία. Είχατε πει, ας πούμε, ότι αν δεν επιτύχουμε κάτι όσον αφορά την προστασία των μητέρων, θα το αποσύρουμε το θέμα. Δηλαδή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάρα πολύ καλό αυτό. Και πιστεύω ότι θα το κάνατε. Τι έγινε. Συγγνώμη, υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο του μιλητή. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα σημαντικά θέματα της Ευρώπης. Έχω δύο ερωτήσεις. μία αφορά το πρόγραμμα Juncker. Στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή συζητείται το γιατί αυτά τα κονδύλια τα οποία θα προσφέρουν εγγύηση γιατί αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να προέρχονται από τον τομέα της έρευνας. Γιατί λοιπόν δεν συμμετέχουν περισσότερο, γιατί δεν επιβαρύνονται περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία. Μήπως ήταν σκόπιμο στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης να διαμορφωθούν διαφορετικά ε, τα ε, χρηματοδοτικά κονδύλια, δηλαδή πρόγραμμα Juncker και συμπληρωματική χρηματοδότηση. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά το Better Regulation. Εσείς ε, είπατε ότι θέλετε να καταπολεμήσετε περισσότερο τη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία και είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όργανο που να παρεμβάλλεται ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Νομίζω ότι και εμεί το ζητήσαμε αυτό στο ψηφισμά μας ε, του Νοεμβρίου στο άρθρο 21. Αναφέρεται αυτό. Όμως το ερώτημα που τίθεται τώρα, μέχρι ποιου σημείου θα υπάρχει ανεξαρτησία από την Κομισιόν. Ε, το δεσμευτικό τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέχρι ποιο σημείο φτάνει και αυτό. Επιτρέπεται ο έλεγχος της επικουρικότητας και μέχρι ποιο σημείο. Στο θέμα αυτό η Ευρώπη είναι ο σωστός νομοθέτης. Αυτό λοιπόν το όργανο που θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στους τρεις θεσμούς, τι ακριβώς αρμοδιότητες θα έχει, αν θέλετε, μέχρι ποιο σημείο θα μπορεί να προχωρήσει. Ο κύριος Μαρτάν εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο, θα είμαι σύντομος. Είπατε πριν από λίγο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προτεραιότητα της Επιτροπής και συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως πάνω σε αυτό να σας επισημάνω ότι υπάρχει ένας τομέας ο οποίος έχει υποφέρει πολύ τα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή ε, ενέργειας ή μάλλον η παραγωγή φωτοβολταϊκών η Κίνα έχει κατακλείσει την ε, αγορά με τα δικά της φωτοβολταϊκά. Το ερώτημα τώρα, εάν ήταν ε, λάθος της Ευρώπης, πρέπει να μας προβληματίσει, αλλά πίσω από αυτή την κίνηση είναι, ε, βρίσκεται και το ίδιο το κράτος, το ίδια η Κίνα. Γιατί η Κίνα έχει δώσει κρατικές ενισχύσεις στις εταιρείες της που παράγουν φωτοβολταϊκά. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι πιστεύετε γι' αυτό, μήπως σε, κάποιες, ε, σε κάποιους τομείς της βιομηχανίας, τους οποίους ε, αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις, τέτοιους κινδύνους από το τρίτες χώρες, πώς θα πρέπει να αντιδρούμε. Πώς θα πρέπει να αντιδρούμε όταν υπάρχει μια χώρα η οποία προσπαθεί να ε, επέμβει στην οικονομία την ευρωπαϊκή. οι ευρωπαϊκές συνθήκες ε, διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό και ε, την, ότι δεν θα υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Και όσον αφορά λοιπόν την πολιτική μας για την ανακύκλωση και για τα απορρίμματα, η πολιτική, η, τακτική ορισμένων κινέζικων εταιριών μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό, για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, όταν η Ευρώπη έχει κάποιου κανόνες για την ασφάλεια για παράδειγμα και του επιβάλλει, δε, δεν θα έπρεπε κατά αντίστοιχο τρόπο να έχουμε επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων και σε αυτά τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά. Με αυτόν τον τρόπο μάλιστα θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε και να, να, να ενθαρρύνουμε και τις άλλες χώρες, τις άλλες υπήρους να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για τους συντηρητικού κύριο Ντάνκαν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σας μιλήσω σύντομα για το ε, πλέγμα της Βόρειας ε, Θάλασσας. Προχωρούμε με την αξιολόγηση αντικτύπου. Ωστόσο, κατά το παρελθόν έχουμε διαπιστώσει ότι είχαν γίνει αξιολογήσεις αντικτύπου που δεν ήταν ε, κατάλληλε, δεν, ήταν οι απαιτούμενε, δεν είχαν την απαιτούμενη ποιότητα. Και μας ενισχύει λίγο η κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει αυτή η νομοθεσία. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Βόρεια Θάλασσα, τα οποία θα ήθελαν η αξιολόγηση αντικτύπου να, γίνει, να είναι υψηλή ποιότητας και εύλογη και λογική, τότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο και να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε για το ενεργειακό πλέγμα στην περιοχή αυτή, το οποίο είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια συνολικά. Αυτό όμως περνάει από την σωστή αξιολόγηση αντικτύπου. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνκαν. Εκ μέρου του Άλντε. Κύριε Σέντερλε. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα που σας είχα θέσει και όταν ε, συζητήσαμε στην ε, συνεδρίαση της ομάδας Άλντε. Υπάρχει το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας, γιατί μπορεί να ψηφίζεται ε, ορθή ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην υλοποιείται σωστά στα εθνικά κρατημέλη ή ακόμα χειρότερα να μην υπάρχουν κατάλληλοι ελεκτικοί μηχανισμοί. Με άλλα λόγια, πώς θα κτίσουμε μηχανισμούς στην Ευρώπη που θα διασφαλίζουν την ε, εμπιστοσύνη. Πολύ συχνά έχει διαπιστωθεί το φαινόμενο οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι ορθέ, αλλά να μην εφαρμόζονται σωστά, να μην μεταγράφονται σωστά στο εθνικό δίκαιο των διαφόρων κρατών μελών. Και το ένα ζήτημα είναι η μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο, στην εθνική νομοθεσία, και το άλλο ε, είναι ο τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον τρόπο να τιμωρούμε, ή εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε πρόστιμα ή κάτι, κάποια άλλη μορφή, έτσι ώστε να, να, να διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία υλοποιείται στην πράξη. Ξέρω ότι οι απόψει μου δεν, είναι, δεν θα ήταν και τόσο δημοφιλεί στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει να έχουμε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει εκείνη από την πλευρά τη, έτσι ώστε αυτά που λέμε σε αυτό το κοινοβούλιο να, να, να εφαρμόζονται στην πράξη. Κύριε Σιλικιώτη. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, εγώ θα πάω σε ένα άλλο θέμα ε, και αναφέρομαι στις διαδικασίες που εφαρμόζει η Τρόικα μέρος της οποίας είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα μνημόνια. Στην έκθεση που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τον ρόλο της Τρόικας τονίζονται πως τα σκληρά μέτρα λιτότητας παραβιάζουν τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν συμβαδίζουν με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γίνεται δε κριτική ότι τα μνημόνια δεν λαμβάνουν υπόψη του τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν ω αποτέλεσμα να ανοίγει η ψαλίδα κατανομή του πλούτου, να διευρύνονται οι κοινωνικέ ανισότητε, η ανεργία να καλπάζει στα ύψη, ειδικότερα μεταξύ των νέων. Εσεί πώ αξιολογείτε μέχρι στιγμή την εφαρμογή των μνημονίων στα κράτη-μέλη, από αυτήν τη σκοπιά, δηλαδή από τη σκοπιά τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι θα πράξετε ε, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βγάζουν από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την λήψη των αποφάσεων, ποια μέτρα θα προωθήσετε ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία. Και ε, επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι πώς θα διασφαλιστεί ότι μέσα από κανονισμούς να περιορίζεται η αδιαφάνεια που υπάρχει στη δράση των διαφόρων ομάδων, κυρίως οίκων οι οποίοι ασκούν διάφορες πιέσεις συγκεκριμένα ε, για να προωθήσουν συγκεκριμένα εταιρικά συμφέροντα. Και το λέω αυτό διότι παραβιάζεται μια βασική αρχή με τη δράση αυτών των οίκων του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. On behalf of e Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορέλη από το EFTD. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Όπως σας έχω ήδη πει στη διάσκεψη των Προέδρων, ε, συνήθως κρίνω τα αποτελέσματα και ποτέ τις προθέσεις. Επομένως, ευπρόσδεκτη αυτή η νέα μέθοδος εργασίας. Αν μας οδηγήσει στα προσδοκόμενα αποτελέσματα, θα είμαι ο πρώτος που θα σας χειροκροτήσω. Θυμάμαι όμως ότι τότε είπατε ότι ε, βγάζουμε από την συζήτηση πολλά θέματα τα οποία ήταν αρκετά παλιά. Και είδα και το θέμα της κυκλικής οικονομίας το οποίο αποσύρθηκε, ενώ εσείς λέτε τώρα ότι θα το επανεισάγετε. Δεν καταλαβαίνω το εξής. Επειδή ακριβώς ε, είχε λιγότερο από ένα χρόνο ζωή. Θα ήθελα να ξέρω καταρχά πότε ακριβώ θα το επανεισάγετε, διότι θεωρώ ότι όπω και εσεί ε, θεωρούμε ότι η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει ε, μεγάλο ε, και η καταπολέμησή τη σημείο όφηση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και θα ήθελα να ξέρω τι διαφορετικό υπάρχει σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση για να δικαιολογήσουμε και για ποιο λόγο έγινε αλλαγή, που φαντάζομαι ότι γι' αυτό έγινε. Και σα ευχαριστώ και για την απάντησή σα. Ευχαριστώ και να δώσουμε τώρα το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές πέραν των συντονιστών. Η κυρία Τελκαστήγιο έχει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λόγω κάποιων ερωτήσεων που ακούσαμε θα ήθελα να διευκρινίσουμε λίγο ακόμα ε, το λεγόμενο Συμβούλιο Νομοθετικής Εποπτείας, το Legislative Scrutiny Board. Πότε θα μπορέσουμε να καθορίσουμε ή θα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να καθορίσει λίγο σαφέστερα τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτό το ε, πάνελ ε, νομοθετικού ελέγχου. Ε, η πρώτη με ερώτηση λοιπόν είναι λίγο το χρονοδιάγραμμα επ' αυτού και η δεύτερη ερώτησή μου έχει σχέση με αυτή την παρατεταμένη νομοθετική διαδικασία που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που υπάρχει συναπόφαση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ε, μπορεί η μελέτη επιπτώσεων που έχει γίνει αρχικώς ε, να πρέπει να αναθεωρηθεί λόγω της καθυστέρησης. Υπάρχει κάποια πρόγνωση ε, για το τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ε, καλωσορίζουμε κύριε Τίμερμαν, ε, κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω δύο ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν όλοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο θέμα των υπερβολικών νομοθετημάτων, στο θέμα του οικολογικού σχεδισμού, τι θα γίνει στην Κομισιόν, γιατί αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το πώς μπορούμε να τρελάνουμε τους ανθρώπους από το πρωί μέχρι το βράδυ με περιτές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ε, η ε, Κομισιόν λοιπόν θα είναι λιγάκι πιο συνεπής ε, στον περιορισμό όλων αυτών των κανονισμών και κάτι άλλο πάλι για τους κανονισμούς. Εάν θέλουμε να περιορίσουμε τη βιομηχανία στο 20% γιατί επιθυμούμε την οικονομική ανάπτυξη που όλοι τη θέλουμε αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, σκεφτούμε λιγάκι το θέμα των υπερβολικών ρυθμίσεων. Αυτό το 20% ποσοστό βιομηχανίας πώς μπορείτε να το επιδιώξετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ταγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώς λοιπόν σήμερα παρά τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί ε, στην Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στην πρόσβαση στην κοινωνική χρηματοδότηση. Ορίζοντας 2020, πρόγραμμα Κόσμος ή ε, Κόσμε Θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει κάποιο βήμα προς τα εμπρός για να υπάρχει καλύτερη και πιο εύκολη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλα αυτά τα κοινοτικά προγράμματα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν επίτροπος για τις μεταφορές, για μένα τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο ε, να εφαρμόσω το πρόγραμμα Μαρκο Πόλο. Πολλές δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις γιατί ήταν πάρα πολύ ε, περίπλοκο το θέμα. Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σορίνιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ε, πω ότι η καλύτερη νομοθεσία είναι μια πολύ καλή διαδικασία που αφορά στην ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια κάτω από το πρίσμα το ότι υπάρχει μια παγκόσμια πλέον οικονομία. Το θέμα είναι, ή το θέμα, το πρόβλημα δεν έχει σχέση με την νομοθεσία, αλλά με το επίθετο καλύτερη. Εάν λοιπόν εκφράσουμε όλοι μας την απόψή μας, θα δούμε ότι ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία στο ότι είναι καλύτερη νομοθεσία και τι θέλει κανείς να πετύχει. Για μένα, παραδείγματος χάρη, στην ενέργεια καλύτερη νομοθεσία σημαίνει καλύτερη ή μεγαλύτερη επάρκεια, καλύτερη χρήση των πόρων, επάρκεια ε, πόρων στις οικονομίες μας. Σημαίνει επίσης λιγότερο επιθετική προσέγγιση στην οικονομία και στο περιβάλλον. Και υπάρχει και ο ψηφιακός τομέας. Όλοι μας έχουμε κατά νου το ότι πρέπει να είναι η ψηφιακή οικονομία, κατόπιν υπάρχουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και εκεί δεν ξέρω τι ερμηνεία μπορεί κανείς να δώσει και υπάρχουν και οι ρυθμίσεις ε, για τους φορολογικούς παραδείσους, ε, για τις ε, κρατικές προμήθειες, δημόσιους διαγωνισμούς. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι η καλύτερη νομοθεσία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά πρέπει να έχουμε ένα όραμα το οποίο θα δημιουργεί κάποια εξέλιξη. Εντάξει, να υπάρχει κάποια κατεύθυνση πολιτικής, αλλά το ζητούμενο είναι οι πολίτες ε, και νομίζω επ' αυτού καλούμεθα να τοποθετηθούμε. Στις 25 ε, θα έχουμε μία ανακοίνωση για την Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Ε, νομίζω πρέπει να έχουμε πολλές καλύτερες τέτοιου είδους ενώσεις και μετά να προχωρήσουμε στην καλύτερη νομοθεσία. Η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Τίμερμαντ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπω ακούστηκε προηγουμένω, αναφερόμαστε στη μείωση του γραφειοκρατικού άχθου, ιδιαίτερα για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και τη μείωση τη γραφειοκρατία. Ε, ε, αυτό θεωρήσετε ότι είναι προτεραιότητα στη δουλειά σα. Πώ σκοπεύετε όμω να προχωρήσετε σε αυτό το θεματολόγιο για τη μείωση του άκθου. Τι σκοπεύετε να κάνετε από αυτού και ποιο είναι ο τελικό στόχο που θέλετε να επιτύχετε. Και κάτι ακόμα, πώς θα ε, εντάξετε το όλο θέμα αυτό της μείωσης της γραφειοκρατίας με άλλες πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, από τις οποίες ε, θα μπορούν πραγματικά να υποφοληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η αναθεώρηση του Small Business Act δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε ολόκληρη συζήτηση από αυτού πέρσι, έγινε διαβούλευση, πήγατε, πήρατε πάμπολες απαντήσεις. Τι συνέβη λοιπόν με όλα αυτά και πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερπράντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα το απόγευμα. Όπως ε, διαπιστώνετε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τη γραφειοκρατία και κυρίως για το μέγεθος της γραφειοκρατίας. Και αυτό φυσικά δικαιολογείται. Και εγώ συνήθως έχω δύο καλούς κανόνων και έναν κακό κανόνα. Δεν μπορούμε να αναλύουμε τη γραφειοκρατία μόνο από πλευράς ποσότητας, αλλά και από πλευράς ποιότητας. Και εδώ θα έρχεται και το ερώτημά μου. Ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνεται η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τμήμα της ερώτησης. Και η σχέση μεταξύ νομοθεσίας και κανονισμών είναι πολύ σημαντική. Το βασικό ερώτημα λοιπόν εδώ είναι η βασική στάση πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια συλλογή διαφόρων κρατών μελών. Ε, Απλώς ε, η αίσθηση δική μου είναι ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν νιώθουν ότι είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Αναφέρονται στις Βρυξέλλες ως κάποια μακρινή ε, οντότητα στην οποία δεν νιώθουν ότι ανήκουν στην πραγματικότητα. Επομένω, τα πάντα ε, ε, εντάσσονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό έχει και βαθιές συνέπειε στην ποιότητα της νομοθεσίας αν δούμε για παράδειγμα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ή τις μεταρρυθμίσεις της γεωργικής πολιτικής. Η νομοθεσία η οποία εγκρίθηκε ε, πόρο απέχει από τις αρχικές προτάσεις και άλλαξε τόσο πολύ από τα ίδια τα κράτη-μέλη που ε, είναι εκ διαμέτρου διαφορετικοί και πολλές φορές γίνονται για να εξυπηρετήσουν τα ε, εθνικά του συμφέροντα. Αν δείτε το σχέδιο Γιούγκερ, έχουν γίνει ήδη αρκετέ τροπολογίες από τα κρατη και αυτές οι τροπολογίες αντανακλούν τρόπο με τον οποίο θα μπορούν τα κρατη να χρηματοδοτούνται περισσότερο από την Ευρώπη και όχι ε, μια πραγματική απόπειρα να υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι μάλλον το κλειδί του προβλήματος. Το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ιδιαίτερα επικριτικό επ' αυτού ε, συν το χρόνο και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη τη δική σας για τη στάση των κρατών μελών και για το πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Ευχαριστώ κύριο Μπένσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. First of <laughs> uh, Καταρχάς, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Τίμερμαν που ήρθε εδώ σήμερα. Take it's a uh, late payment directive. Έχω μια ερώτηση για την οδηγία για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Αυτό μας δίνει πρόσβαση σε κεφάλαια, σε αγορές και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Η πρόσβαση σε κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό, ε, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την οδηγία για τις κασεμένες πληρωμές και να δούμε ε, αν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ε, γιατί σίγουρα δεν λειτουργεί στη χώρα μου στη Δανία, διότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι μεγάλες επιχειρήσεις, παραδείγματο χάρη αλυσίδες λιανικής, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μικρότερες επιχειρήσεις ως έναν τρόπο να λαμβάνουν πίστοση. Διότι αγοράζουν αγαθά, πολύ συχνά τα πολλούν μέσα σε μερικές ημέρες ε, σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώληση, αλλά αποπληρώνουν τους μικρούς προμηθευτές τους ε, μετά από 60 μέρες. Επομένως, οι μεγαλύτεροι έχουν μόχλευση επί των νεότερων. Τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτό. Η κυρία Βίρκονεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μπορούσα να σας δώσω κίνητρα για να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και να μειώσουμε το άχθος ε, στην Επιτροπή μας. Θα θέλαμε να έχουμε καλύτερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας ε, στην Ευρώπη και γνωρίζουμε ότι για τις επιχειρήσεις μας το πλέον σημαντικό είναι να υπάρχει νομοθεσία και ένα ε, περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και των προτέρων. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλα τα προβλήματα και θα πρέπει να είμαστε δραστήριοι, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του μέλλοντος, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να εργάζονται ε, απρόσκοπτα. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις συνέπειες των εργασιών μας και γνωρίζουμε ότι το σχέδιο επενδύσεων είναι καλό. Ε, τώρα που έχετε αφαιρέσει και 80 διαφορετικά προγράμματα που δεν ήταν και τόσο καλά, γνωρίζω ότι θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στην οδηγία και ε, δεν θα τα προκρίνεται στην αρχική πρόταση. Και έτσι θα πρέπει να γίνει μια νέα αξιολόγηση επιπτώσεων για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή νομοθεσία. Σα εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω πραγματικά να έχουμε βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτό χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Mr. please. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και έρχεστε να μας μιλήσετε για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και δεν περίμενα ότι θα σας έθετα ερώτηση και πάλι, διότι ε, πλέον μετά από όλες αυτές τις συναντήσεις θα πρέπει να δούμε και τι θα έχουμε ως αποτέλεσμα. Ε, αυτό το ανέφερε και ένας από τους συναδέλφους από την ομάδα Στόιμπερ. Μάθαμε ποιες είναι οι προθέσεις σας για αυτό το Συμβούλιο Εποπτείας ε, που θα είναι ένας πιο ανεξάρτητος φορέας και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι έχετε κατά νου. Μετά από 7 χρόνια ε, συμμετοχή σε αυτή την ομάδα Στόιμπερ. Πραγματικά θα ήθελα ε, να αναρωτηθώ αν όντω ήταν ανεξάρτητη, γιατί δεν ήταν. Μπορούσε να θέσει η ίδια το θεματολογιό της. Δεν μπορούσε. Το έθετε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές φορές ε, είχαμε κάποια δυνατότητα να επηρεάσουμε και εμεί λόγω των διαβουλεύσεων. Ουσιαστικά η γραμματεία μας ήταν υπάλληλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαμε ίσως να ε, χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας για να αντιτάξουμε κάτι στις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούσαμε γιατί δεν είχαμε δικό μας προπολογισμό και δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη. Επομένως θα ήθελα να ξέρω... Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το σύστημα, θα υπάρξει μια δέσμη προτάσεων και θα πρέπει να το αναλύσουμε μαζί σας και ίσως να υπάρξει και κάτι από πλευράς μας. Αλλά όσον αφορά την ανεξαρτησία, και τον ίδιο αυτό το φορέα, αυτό το συμβούλιο, θα μπορούσατε να μας δώσετε μια μικρή γεύση του τι ακριβώς αναμένετε ότι θα είναι αυτό το συμβούλιο, τι καθήκοντα θα έχει και τι υπηρεσίες θα παρέχει. Ευχαριστώ. Και τέλος, τελευταίο στον κατάλογο, πριν ε, λάβουμε όλες τις απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις, ο κύριος ε, Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ένας φίλος μου επιχειρηματίας πριν από κάποια χρόνια, όταν τον ρώτησα, γιατί τότε εγώ άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ω πολιτικοί για να σας βοηθήσουμε. Και η απάντησή του ήταν, καταρχάς, ίσως για έξι μήνες να μην αποφασίσετε τίποτα καινούργια. Καμία νέα νομοθεσία, κανένα νέο κανονισμό. Μου φάνηκε πολύ καλή απάντηση. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Έσπα μια ιστορία σας λέω εδώ. Αλλά πριν αρχίσω να ασχολούμαι με την πολιτική, και εγώ ήμουνα ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης και αντιλαμβάνομαι ότι μία από τις δυσκολίες ε, του να είναι κάποιος επιχειρηματίας είναι το να συμμορφούνται με όλη την ομοθεσία η οποία τίνει να αυξάνεται και ποτέ να μειώνεται. Αυτή είναι και η δυσκολία. Είναι μία μηχανή που συνεχώς ε, τροφοδοτείται. Κατά την άποψή σας κύριε Αντιπρόεδρε, Ποιος είναι ο ρόλος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσει το γεγονός αυτό, διότι ε, κάποιο τμήμα αυτής της νομοθεσίας είναι εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ίσως μπορεί να είναι και κακή ή ελλειπώς σχεδιασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας, κάποια είναι πρωτότυπη εθνική νομοθεσία, υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες και στην εθνική νομοθεσία και τι είναι αυτό που κατά την άποψή σας ε, θα μπορούσατε να κάνετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να φτάσουμε πραγματικά στο επίπεδο όπου το 90 ε, τόσο που εργάζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς. Παρακαλώ έχετε το λόγο πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα να μας πείτε. Παρακαλώ. Indeed. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες όσο καλύτερα μπορώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με την σειρά που ετέθησαν τα ερωτήματα αλλά ίσως ομαδοποιήσω και κάποια από τα ερωτήματα που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι. Πολλά μέλη του Κοινοβουλίου μάλλον. Πρώτα απ' όλα, για το πρόγραμμα Juncker και το Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και το γεγονός ότι τα κονδύλια από αυτό προέρχονται από ανακατονομή κονδυλίων που αρχικά είχαν προπολογιστεί για τον προπολογισμό της έρευνας. Ειλικρινά, πιστεύω ότι τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την καινοτομία. Αντιθέτως, με αυτό το σύστημα θα δώσουμε τη δυνατότητα ε, πιο εύκολα να υπάρξουν ιδιωτικές επενδύσεις και έτσι να υπάρξουν πιθανότατα και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, περισσότερες από ό,τι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε αν είχαμε μείνει στο πρόγραμμα Horizon 2020. Επίσης, να επισημάνω ότι αυτό το γεωδοτικό ταμείο θα υλοποιηθεί σταδιακά και κατά κύριο λόγο τα κονδύλια έχουν προπολογιστεί για, αργότερα, για, για, για κατοπινές χρονιές. Το οποίο σημαίνει ότι φέτος και την επόμενη χρονιά ε, δεν αναμένουμε μεγάλες ανακατονομές, μεγάλες αλλαγές. Συνολικά, όμως, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα καταφέρει τους τα επόμενα έξι χρόνια να προκαλέσει περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας από ότι αν είχαμε μείνει στο παραδοσιακό σύστημα. Τώρα για τις αξιολογήσεις αντικτύπου και το κατά πόσο αυτές γίνονται με τρόπο αμερόλεπτο, ανεξάρτητο, ένα θέμα που έθεσαν πολλοί βουλευτές. Πρώτα απ' όλα να πω ότι πιστεύω ότι και με το σημερινό καθεστώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις αξιολογήσεις αντικτύπου. Υπάρχει ένα Ε, ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό, να εξασφαλίσουμε ότι εκείνοι οι οποίοι τελικά διεξάγουν την αξιολόγηση αντικτύπου θα έχουν αποδείξει εμπράκτως την ανεξαρτησία τους και όχι απλώς ότι εργάζονται στον τομέα, ότι είναι ειδικοί στον τομέα. Οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι βρίσκονται στο ε, Συμβούλιο Αξιολόγησης των, των αξιολογήσεων αντικτύπου που προετοιμάζουν οι υπηρεσίε τη Επιτροπής. σε ορισμένε περιπτώσει αυτό το Συμβούλιο αναπέμπει αξιολογήσει αντικτύπου στις υπηρεσίε τη Επιτροπής. Εν τέλει όμως, και αυτό το ανέφεραν και ορισμένοι από τους βουλευτέ, η αξιολόγηση του αντικτύπου δεν είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου της πρόταση τη Επιτροπή και μόνο, θα έπρεπε η αξιολόγηση αντικτύπου να ακολουθά την νομοθετική, την ε, νομοθετική διαδικασία. Γιατί αν υπάρξει μια σημαντική μεταβολή στη διάρκεια της διαδικασίας της προτινόμενης νομοθεσίας πρέπει να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το, ποιο θα είναι το αντίκτυπο. Ε, μην ξεκινάμε απλώς με μια αξιολόγηση αντικτύπου η οποία εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής γιατί γνωρίζουμε ότι συχνά κατά τη διάρκεια των ε, μηνών μπορεί η Επιτροπή να έχει προτείνει ενάλογο και με τις αλλαγές που επιφέρει το Συμβούλιο και άλλοι φορείς τελικά να αποκτά μια καμήλα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας αυτήν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και το λέω πολύ προσεκτικά συχνά είμαστε τόσο χαρούμενοι που επιτύχαμε συμβιβασμό που προσπαθούμε να μην τον αγγίξουμε και, προτιμάμε ούτε καν να, αξιολογήσουμε το κατά πόσον αυτός ο συμβιβασμός είναι εφικτό να υλοποιηθεί στα κράτη-μέλη. Πόσο μάλλον τον αντίκτυπο του αυτού, αυτού του συμβιβασμού. Θα ήμουν λοιπόν πολύ χαρούμενος εάν τα κράτη-μέλη συμφωνούσαν να κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου της τελικής νομοθετικής πρότασης, όχι απλώς της πρότασης της Επιτροπής. Και πιστεύω ότι σε αυτό θα συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο γιατί έτσι ενισχύεται η λογοθεσία του Συμβουλίου. Αντιλαμβάνεστε βεβαίω, αντιλαμβανόμαστε βεβαίω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό και δύσκολο πολιτικό ερώτημα, αλλά το ερώτημα είναι το εξή. Έχουμε το θάρρο να αμφισβητήσουμε παλαιότερου συμβιβασμού και να πούμε ότι πρέπει η αξιολόγηση αντικτύπου να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Και πιθανώ να αναθεωρεί και του συμβιβασμού που επιτυχάνονται μεταξύ συμβουλίου, στο Συμβουλίο. Εάν και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνήσουν και τα τρία, όχι μόνο η Επιτροπή, και τα τρία συμφωνήσουν ότι θα έχουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου από την αρχή ως το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή δεν θα αντιταχθεί αντι, αντι, Αντιθέτω, εμεί θα υποστηρίξουμε ένα πλήρω αμερόληπτο, ένα πλήρω ανεξάρτητο Συμβούλιο Αξιολόγηση Αντικτύπου. Με την προϋπόθεση όμως ότι και τα τρία θεσμικά όργανα θα συμφωνήσουν ότι θα υποβάλουν τις προτάσεις τους, τι θέσει τους σε ένα τέτοιο συμβούλιο. Μα δώσατε το παράδειγμα της Δανίας, όπου υπάρχει ένα συμβούλιο που γνωμοδοτεί και μετά οι νομοθετικέ αρχές ε, είτε ακολουθούν την εισήγηση είτε ε, αιτιολογούν γιατί δεν, το, δεν ακολούθησαν την εισήγηση. Πάντω, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα που θα το θεωρούσα ιδανικό, πρέπει να συμφωνήσουν και τα τρία θεσμικά όργανα, όχι μόνο η Επιτροπή. Είναι όμω ένα ζήτημα εξαιρετικά περίπλοκο σε πολιτικό επίπεδο για να βρεθεί μια συμφωνία εδώ. Εάν όμω και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνήσουν ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα τη νομοθεσία, να φτάσουμε σε νομοθεσία η οποία θα μπορεί να εφαρμόζεται καλύτερα στα κράτη-μέλη, αν είμαστε ε, ειλικρινεί ω προ αυτήν την πρόθεση, πρέπει να φτάσουμε σε μια αξιολόγηση που η οποία να αξιολογεί την νομοθετική πρόταση όπω αυτή διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου και όχι μόνο αυτό που αρχικά πρότεινε η Επιτροπή. Και επίσης είναι σημαντικό το ζήτημα της ανεξαρτησίας, της ημεροληψία. Είναι κάτι το οποίο το, το επισημούν και τα τρία όργανα πιστεύω. Να το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι και τόσο δίκαιο ένα μόνο από τα τρία θεσμικά όργανα να υπόκειται σε ανεξάρτητο ε, ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση ενδεικτύπου και τα άλλα δύο να μπορούν να ανοίξουν τα σχήρα τους, πρέπει να βρεθεί καλύτερη ισορροπία. Τώρα στο ζήτημα των εμπορικών πρακτικών που έθεξε ο κύριος Μαχτά. Είναι ένα ζήτημα περίπλοκο και πολύ σημαντικό βέβαια. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες κατά του dumping για την επίλυση συγκρούσεων κτλ. Ωστόσο, πολλές φορές η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η πραγματική οικονομία ξεπερνά τους κανόνες. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο γρήγορα θα έπρεπε με το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχω σήμερα να σας δώσω μια συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα που αναδείξατε. Πάντως, σήμερα να σας πω ότι συναντήθηκα με προσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Χαλιβουργίας, οι οποίοι μου εξήγησαν ότι αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό από την Κίνα, που προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, για να το θέσω ευγενικά, και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα στο υφιστάμενο σύστημα. Και πιστεύω ότι και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Μάλλον αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί στο, στα φόρα του ε, Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Χωρίς λοιπόν να έχω μια συγκεκριμένη λύση να σας προτείνω, τουλάχιστον να σας πω ότι η θέση μου είναι ότι ο προστατευτισμός σε κάθε περίπτωση είναι απευκταίως θα ήταν η χειρότερη δυνατή λύση, αν και δεν πιστεύω ότι ο κ. Μαχτάν θα ε, υποστήριζε τον προστατευτισμό. Σε αυτό σίγουρα συμφωνούμε, τουλάχιστον οι δυο μας. Αλλά ένα πράγμα που έμαθα από την εμπειρία μου στα ζητήματα της ενιαίας αγοράς είναι ότι όταν η Ευρώπη αποφάσισε με τον Τελόρ να δημιουργήσει αυτή την ενιαία αγορά με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασκήθηκε κριτική από διάφορους κλάδους της οικονομίας, κλάδους της βιομηχανίας στην Ευρώπη, τότε ήδη, που έλεγαν ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παγκοσμίω εάν ε, θέσουμε υψηλά πρότυπα. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι τόσο σημαντική που εάν τα πρότυπα αναβαθμιστούν στην Ευρώπη, οι υπόλοιποι παίκτε στον κόσμο, επειδή θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, σιγά σιγά ευθυγραμμίζονται. Επομένως, δεν συμφωνώ με τη λογική που λέει ότι όταν αυξάνουμε, όταν ε, βελτιώνουμε τα πρότυπα ποιότητα στην Ευρώπη, αυτό μας καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς. Έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό τα τελευταία χρόνια, τα, τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε καταφέρει να επιβάλλουμε υψηλότερα πρότυπα ποιότητα στην Ευρώπη. Για τον κύριο Ντάνκαν, για το ενεργειακό, για το ηλεκτρικό ε, δίκτυο ε, της Βόρειας Θάλασσας. Όσον από την πλευρά της Επιτροπής μπορώ να σας πω ότι η Ενεργειακή Ένωση και η διασύνδεση είναι πρώτης προτεραιότητας. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει όταν διαπίστωσα πόσο μεγάλα προβλήματα διασυνδεσιμότητας υπάρχουν στις, στις, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα παραγωγή, ε, μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι κρίμα που υπήρξε περικοπή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το πρόγραμμα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι ο αρμόδιος επίτροπος θα προσπαθήσει να βρει τα απαιτούμενα χρήματα. Πάντως η διασυνδεσιμότητα στην, ε, των ενεργειακών δικτύων θα είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένα θέμα επίσης για, οποίο, το οποίο έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους και πολλοί ιδιώτες επενδυτές. Βεβαίω και θα γίνει η αξιολόγηση που Τώρα δεν καταλαβαίνω. Το, ερώτημα υπονοούσε ότι θέλετε να συζητήσουμε το ζήτημα του φράκινγκ. Αν αυτό ήταν το θέμα, πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρούμε ότι δύο απαιτήσει που πρέπει να υφίστανται για να υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχει προστιθέμενη αξία και να μπορεί αυτό να γίνει καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το εθνικό επίπεδο, καμία από αυτές τις δύο προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την υδρορογμάτωση, το fracking. Τώρα, για τον κύριο Φέντερλι που με ρώτησε για την υλοποίηση της ψηφιστής σας νομοθεσίας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κέριο ερώτημα. Νομίζω ότι εν μέρει οφείλεται στην οικονομική κρίση το γεγονό ότι η παρακολούθηση, η λογοδοσία για το κατά πόσο τα κρατημέλη εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο θα θέλαμε τα τελευταία χρόνια. Η Επιτροπή εντέλεται από τις συνθήκες να παρακολουθεί και να ε, εξασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την ε, νομοθεσία που συμφωνείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό στον τομέα του ανταγωνισμού, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας, να ξεκινούμε διαδικασίες επί παραβάση, αν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να ε, πείσουμε, να, να αναγκάσουμε τα κρατη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, την οικονομία των κρατών μελών και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετέφει επίσης ένα ερώτημα για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων της Τρόικας. Είναι ένα ερώτημα που έρχεται και ξανάρχεται. Δυστυχώς ο κ. Ηλικιώτης που το έθεσε δεν είναι πια στην αίθουσα. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω, θα δώσω την απάντηση που είχα δώσει και στο παρελθόν. Ότι σε μεγάλο βαθμό εδώ είναι ζήτημα του κάθε κράτους μέλους. Αυτή τη στιγμή σε ένα κράτος μέλος συνάπτει μια συμφωνία με την Τρόικα. Και το πιστεύω και γενικότερα αυτό για το μέλλον. Είναι κάτι που έχει ε, αναφέρει και ο πρόεδρος Γιούνκερ πολλές φορές ότι οποτεδήποτε υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, οποτεδήποτε αξιολογούμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, θα πρέπει να υπάρχει και μια αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου. Η αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου πρέπει να είναι μέρο τη αξιολόγηση αντικτύπου τη γενική. Ο κ. Μπορέλη με ρώτησε για το ζήτημα τη Κυκλική ε, οικονομία ε, και τη διαχείριση απορριμμάτων. Και γιατί αυτή την πρόταση την αποσύρουμε. Γιατί πιστεύω ότι είναι ζήτημα ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει υποβάλει προτάσει υψηλότερη ποιότητα. Και σα το λέω αυτό με την ιδιότητά μου ω ε, αντιπρόεδρο αρμόδιο για την βελτίωση τη ποιότητα τη νομοθεσία. Υπάρχει ένα ζήτημα ποιότητα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ο τίτλο ανέφερε μιλούσε για κυκλική οικονομία. Ενώ στην πραγματικότητα μιλούσαμε για απορρίμματα. Λάθο. Το ζήτημα τη κυκλικό οικονομία είναι πολύ ευρύτερο. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πρόταση που να καλύπτει πλήρω την κυκλική οικονομία, δηλαδή πώ ξεκινά ο κύκλο ζωή στην οικονομία αφενό και αφετέρου πώ μπορούμε να, αξιολογήσουμε την ανα... Ε, να αξιοποιήσουμε την ανακύκλωση. Πρόκειται για ιδέες οι οποίες κυκλοφορούν από το 1970. Τι γίνεται από με την παρακολούθηση της ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση, για παράδειγμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση άργησε να υιοθετήσει αυτές τις αναλύσεις, αυτές τις ιδέες, αυτές τις πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω ακόμα και σε σχέση με χώρες όπως η Κίνα σε ζητήματα κυκλικής οικονομίας. Με... Ρωτήσατε κύριε Μπορέλη πότε θα το κάνουμε αυτό. Φέτος σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να χάσουμε την ε, ταχύτητα που είχαμε αποκτήσει. Τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, είχε, προταθεί, είχε υποβληθεί αυτή η πρόταση για τα απορρίμματα ε, δεδομένου ότι δεν ξεκίνησε καν εξέταση στο Συμβουλίο και το Κοινοβουλίο, νομίζω ότι αν υποβάλει μια νέα πρόταση τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο στην πραγματικότητα. Πάντω, επαναλαμβάνω ότι αυτό το πακέτο μέτρων για τα απορρίμματα ε, ε, δεν ήταν επαρκέ αφενό για λόγου ποιότητα τη νομοθετική πρόταση και εξωτερού γιατί δεν κάλυπτε πλήρω τα ζητήματα τη οικονομία. Γι' αυτό το Συμβούλιο Υποπτία και την αξιολόγηση επιπτώσεων και πότε θα πρέπει να γίνει. Υπάρχει κάποιε ερωτήσει του κυρίου Στόιμπερ για την, για... Μάλλον, για την ομάδα Στόιμπερ. Ο κύριος Τελίτσια ρώτησε και αυτός για την ομάδα Στόιμπερ. Θέλω να είμαι πολύ σαφή από αυτού. Το πρόβλημα με την ομάδα Στόιμπερ δεν ήταν το γεγονό ότι η γραμματεία ήταν μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονό ήταν ότι η ομάδα Στόιμπερ δεν είχε ομόφωνη άποψη και τελικώ διαλύθηκε η ομάδα Στόιμπερ. Και θέλω να είμαι βέβαιο ότι όλοι όσοι έχουν κάτι να χάσουν και του ενδιαφέρει καλύτερη νομοθεσία θα πρέπει να έχουν άποψη. Λυπάμαι για παράδειγμα που τα συνδικάτα δεν θεωρούν ότι εκπροσωπούνται από την ε, τελική έκθεση. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον επ' αυτού, θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να προσπαθήσουμε να έχουμε και την άποψή τους για συμπεράσματα και να υποστηριχτούν αυτά τα συμπεράσματα. Και πιστεύω ότι ο κύριος Στόιμπερ έχει πολλά να προσθέσει σε αυτή τη συζήτηση, γι' αυτό και του ζητήθηκε τώρα να είναι ειδικό σύμβουλο ε, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για μένα και θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά και την εμπειρογνωμοσύνη του και την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει τα τελευταία ένα-δύο χρόνια για να βελτιώσουμε με τι προσπάθειε μα σε θέματα ε, βελτίωση τη νομοθεσία. Σίγουρα δεν θα χαθεί η εμπειρογνωμοσύνη του, θα αντλήσουμε από αυτή την εμπειρογνωμοσύνη και θέλω και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπω για παράδειγμα περιβαλλοντικά κινήματα, συνδικαλιστικά σωματεία, να ε, εισακουστούν και αυτοί και να ε, συνεισφέρουν στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να το αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονο ότι όλοι εμεί, όλα τα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό και σε απάντησε και στον κύριο Κάρενς, ο οποίο ε, με ρώτησε από αυτού, ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια εσωτερική αναζήτηση εμεί ω θεσμικά όργανα για το πώ ακριβώ εργαζόμαστε. Κάποιο συνάδελφό σα, δικαίω μα είπε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί στη δημιουργία νέα νομοθεσίας. Αλλά ε, αφιερώνουμε κάποιο χρόνο να εξετάσουμε την προηγούμενη νομοθεσία και να δούμε πώς ε, προχωρά από πλευράς ποιότητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα με τους πολιτικούς σε όλα τα επίπεδα. Και με μένα. Θέλουμε να κάνουμε νέα πράγματα, καλύτερα πράγματα, αλλά ορισμένε φορέ θα πρέπει να μπούμε στον κόπο να δούμε τι κάναμε στο παρελθόν και αν όντω αυτό ε, ε, επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Πρέπει αυτό να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ορισμένε φορέ σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού. Ε, έχω μεταβεί σε αρκετά κράτη-μέλη τι τελευταίε ε, μια-δύο εβδομάδε να μιλήσω απευθεία με επιχειρήσει, κυρίω μικρομεσαίε επιχειρήσει και έμαθα ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλο τους μεγάλους κλάδους να εισακουστούν σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να εισακουστούν εδώ. Δεύτερον, είναι πολύ πιο εύκολο για τους μεγάλες επιχειρήσεις να ε, φροντίσουν να προσαρμοστούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία από ό,τι πολύ συχνά συμβαίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει ε, αυτό το λεγόμενο ε, gold plating, υπερβολική νομοθεσία και κανονισμοί στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές η ευρωπαϊκή νομοθεσία χρησιμοποιείται ως πρόσθετο σε εθνικό, στο εθνικό επίπεδο και ορισμένες φορές στο ε, κατώτερο επίπεδο του εθνικού, σε περιφερειακό και τοπικό. Και αυτό φυσικά είναι πολύ μεγάλος βραχνάς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε καλύτερη νομοθεσία, παρεπιπτόντως αυτός ο τίτλος καλύτερη νομοθεσία δεν καταλαβαίνω προστή, ε, δηλαδή ποιος θέλει χειρότερη νομοθεσία. Ε, δεν είναι και η σούπερ καινοτομία, αλλά το θέμα είναι πώ θα μπορέσουμε να έχουμε καινοτομία. Και αυτή είναι η καλύτερη νομοθεσία και αυτή είναι η καινοτομία μα. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται κεντρικά από τι Βρυξέλλες, θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο πρωτεύουσα και θα πρέπει να υπάρχει και άμεση συμμετοχή των κλάδων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, Και θεωρώ ότι εδώ οι συνήθειες ε, των ε, θεσμικών οργάνων μας είναι να νομοθετούμε. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα θα σας προτείνουμε μια νέα πρόταση για οδηγία και εσείς αποφασίζετε από αυτή. Αυτός είναι ο συνήθις τρόπος με τον οποίο προχωρούμε. Ε, ε μπορεί να ακούγουμε λίγο επαναστατικός, αλλά μπορεί να μην είναι πάντα η λύση, η νομοθεσία στα προβλήματα όλων και ίσως θα έπρεπε να το εξετάσουμε ε, με λίγο πιο πολιτικό τρόπο. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας ακριβώς ε, και μόνον ελέγχοντας την κείμενη νομοθεσία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπήρξε τόσο πολύ μεγάλη υποστήριξη και στη Μαδρίτη και στο Παρίσι και είμαι βέβαιος ότι θα την έχω και αύριο στο Βερολίνο και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια μεγαλύτερη αίσθηση συνενοχής σε όλα τα επίπεδα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό και σε περιφερειακό ώστε να φροντίσουμε πραγματικά να έχουμε και αποτελέσματα από αυτού. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη ήταν από τους μεγαλύτερους υποστηριχτές ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και τους έχουμε χάσει πλήρως στο ευρωπαϊκό ε, οικοδόμημα διότι δεν βλέπουν πρόοδο, δεν θεωρούν ότι έχουν γίνει και πολλά πράγματα και δεν θεωρούν ότι πρέπει να πλήττονται οι ίδιοι από τις ε, πολύ επαχθείς ε, προϋποθέσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ορισμένες φορές λοιπόν ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό πάρα πολύ προσεκτικά διότι πλέον δεν είναι με το μέρος μας. Τώρα, οικολογικός σχεδιασμός Δεν έχω εδώ κάποια ρηξικέλευτη δήλωση σαν αυτή του κυρίου Ρόιλ για τον οικολογικό σχεδιασμό εν γέννη. Θεωρώ ότι είχε κάποιες πολύ θετικές συνέπειες, κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση. Και αν ε, θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία, πρέπει να μειώσουμε ουσιαστικά την ενεργειακή μας κατανάλωση. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό ε, με την ομοθεσία για τη βιομηχανία που θα απαιτεί οι ηλεκτρικές συσκευές να κλείνουν αυτόματα μετά από ε, μια περίοδο αδράνειας. Όλοι ξεχνάμε να κλείσουμε μια ηλεκτρική συσκευή. Αν κλείνει αυτομάτως, ε, τότε αυτόματα ε, είναι ένα μέτρο που μας βοηθάει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Σε γενικές γραμμές ο οικολογικός σχεδιασμός δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι ούτε κάτι καλό. Τα κατάλληλα μέτρα στον οικολογικό σχεδιασμό θα έχουν καλά αποτελέσματα, κάποια άλλα όχι και θεωρώ ότι θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά ένα προς ένα για να είμαστε βέβαιοι ποιο έχει αποτελέσματα και ποιο όχι. Ε, βιομηχανική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικαιρό ζήτημα και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο για το μέλλον της απασχόλησης και της οικονομίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ, πιστεύω ακράδαντα και εδώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα επανεβιομηχάνηση η οποία θα είναι βιώσιμη και θα ε, πηγαίνει ε, προς την άγουσα που θα προοδεύσει και η παγκόσμια οικονομία την επόμενη δεκαετία. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την καινοτομία, αλλά να την ε, εντάξουμε ταυτόχρονα με την ανάπτυξη και την παραγωγή στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι υπάρχει πλέον προσέγγιση των αγορών, επιτροπή ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, που είχε παραδοσιακά απομακρυνθεί και θα πρέπει να είμαστε υπέρ αυτών που δίνουν κίνητρα για αυτές τις εξελίξεις και αν εξετάσουμε τα διάφορα στοιχεία του σχεδίου Γιούνκερ και διάφορους άλλους τομείς, για παράδειγμα ψηφιακή έννοια αγορά, ενεργειακή ένωση και το καθεξής, όλα αυτά αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της εξέλιξης αυτής. Πιστεύω επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εκεί έγκυται και η απασχόληση, η απασχόληση σε όλα τα επίπεδα. Μία από τι μεγαλύτερε αδυναμίε μα στην οποία πραγματικά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή και εθνική δράση, είναι το γεγονό ότι οι δεξιότητε που χρειάζονται και οι δεξιότητε που διαθέτουν οι νεότερες γενιές μα δεν έχουν μια αντιστοιχία. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψη δεξιοτήτων ή κακή αντιστοίχησης δεξιοτήτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική που έχει σημασία για μια βιώσιμη οικονομία, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δεξιότητες που έχουν ε, οι άνθρωποι είναι αντίστοιχες αυτών που απαιτούν ε, οι κλάδοι. Ε, και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε δράση σε όλα τα επίπεδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Ταγιάννη με ρώτησε για τη χρηματοδότηση στην, σε ευρωπαϊκό επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρω ότι η Επίτροπος Μπιανκόφσκα ασχολείται με το θέμα αυτό και έχω τις ίδιες ε, παρατηρήσεις και τα ίδια σχόλια όπου πάω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε να συμμετέχουμε στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά οι κανόνες είναι τόσο περίπλοκοι που ε, χρειάζεται πλήρες ε, νομικός σύμβουλος, σχεδόν ολόκληρο νομικό γραφείο στην επιχείρησή σου για να μπορέσει να υποβάλεις αίτηση για χρηματοδότηση. Και η Επίτροπος Μπιανκόφσκα ασχολείται με το θέμα αυτό νομίζω. Όσον αφορά το Small Business Act, Νομίζω θα έχετε ακούσει από μένα ότι πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται υποστήριξη διότι τόσο το πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και η λύση του έγκυται στο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό κομμάτι των επενδυτικών προγραμμάτων. Και όπως σας είπα, η Επίτροπος Μπινκόφσκα δουλεύει πάνω στη βελτίωση της καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, πρόσβασή του στις παγκόσμιες αγορές, ε, στην ε, καινοτομία και όπως σας είπα και σε εξειδικευμένου εργαζόμενους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει περιορισμό του διοικητικού άχθους και συμφωνώ απόλυτα με τις εθνικές αρχές που θέλουν να το πράξουν αυτό, να το εφαρμόσουν στην πράξη, θα τι στηρίξω ανεπιφύλακτα. Ρίχνω έτσι μια ματιά στις σημειώσεις μου. Νομίζω ότι απάντησα σχετικά με την Ευρωδοσία. Μισό λεπτό, κύριος ε, Χεμπράντη ε, ρώτησε για την στάση των κρατών μελών. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις του επ' αυτού. Η δική μου εμπειρία σε αντίθεση με αυτό που πολλοί πιστεύουν είναι ότι τους τελευταίους τρεις ε, μήνες έχουν εγερθεί υπερβολικές προσδοκίες από πλευράς κρατών μελών απέναντι στην Κομισιόν. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν φοβάμαι αυτές τις ε, προσδοκίες. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα βαρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι οι προσδοκίες είναι τόσο μεγάλες που θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Η απάντηση που δίνω στα κράτη-μέλη είναι ότι θα μπορέσουμε εάν υπάρξει ουσιαστική συνεργασία και αν αυτή η παραδοσιακή ε, πρακτική είναι ότι ό,τι κάνουμε εμείς είναι καλό και ότι κάνουν Βρυξέλλες είναι κακό. Αν το ξεφορτωθούμε αυτό, αυτή τη νοτροπία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λίγο πολύ αυτά είχα να σας πω. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Τίμερμανς, ο κύριος Τσελίτσκα. Έχετε ένα διαδικαστικό, σύντομα παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Είπατε για το πρόβλημα της ομάδας Στόιμπερ ότι δεν εισακούαταν η φωνή των συνδικάτων. Αυτό δεν ισχύει. Μετά από 7 χρόνια που ήμουνα μέλος, το πρόβλημα το βλέπω τελείως διαφορετικά. Με την έννοια ότι η ομάδα δεν μπορούσε να έχει τη δική της, το δικό της αιματολόγιο, απόλυτα εξαρτώμενη από την Επιτροπή που δεν ήθελε αυτή η ομάδα να κάνει καλή δουλειά και καμία πληροφορία δεν μπορούσε να διασταυρωθεί, δεν υπήρχε ούτε ηγετική ομάδα, ούτε όρεξη, ούτε θεματολόγιο. Τα συνδικάτα εισακούστηκαν όποτε το επιθυμούσαν. Ήμουνα σε μόνιμη επαφή μαζί τους. Δεν μπορείτε να έχετε μία ομάδα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά μία ομάδα που να ε, μπορεί να ε, πληροφορήσει σωστά την Επιτροπή. Αυτό δεν έχει σχέση με τα συνδικάτα. Αν θέλετε να έχετε μια επαγγελματική ομάδα, ε, απόλυτα εξαρτώμενη, αυτό ε, σημαίνει όμως ότι η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Κοιτάξτε, όποιος ξεκινάει τις παρατηρήσεις του με κάθε σεβασμό, μάλλον τελικά αυτό που κάνει είναι να μην δείχνει κανένα σεβασμό. Η παρατηρήση του κ. Τελίτσκα πράγματι είναι αξιοσέβαστες, δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Δεν είναι ότι δεν ακουγόταν η φωνή τους. Εγώ θέλω να πω ότι οι επιπτώσεις της... Ε, η θετική ενέργεια από την έκθεση αυτή θα μπορούσε να είναι τόσο σημαντική που ε, θα μπορούσε να αξιολογηθεί πολύ καλύτερα. Αυτό ήθελα κατ' ουσία να πω. Είναι πολύ εύκολο να πει κανεί ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν μα άφησε η Επιτροπή για το ένα για το άλλο. Μα η Κομισιόν έδωσε βοήθεια στην ομάδα στο Έμπερ. Τι άλλο να έκανε. Η Κομισιόν, κοιτάξτε, συγγνώμη, με κάθε σεβασμό, αν εσεί σε μία πρόταση λέτε ότι η Κομισιόν ε, προσέφερε τη γραμματεία και μετά λέτε ότι η Κομισιόν ε, δεν προσέφερε υποστήριξη, αυτό δεν είναι συνεπές ως ε, σκέψη Όσον αφορά τον έλεγχο, εγώ λέω ότι ο έλεγχος θα πρέπει να είναι όσο πιο ανεξάρτητος γίνεται. Εγώ θέλω ε, τα, οι εμπειρογραμμονείς να είναι μέλη της ομάδας ελέγχου. Να υπάρχει ισορροπία. Σε 5-6 κράτη-μέλη έχουμε ανεξάρτητα συμβούλια και αυτά μου έχουν συμβουλεύσει και θα το λάβω υπόψη μου ότι στην ισορροπία ισορροπία δυνάμεων στα ελεγκτικά συμβούλια, να είναι ανεξάρτητοι αυτοί, να μην εκπροσωπούν άμεσα τη βιομηχανία τους, ε, τις μονάδες του κράτους τους. Κύριε Σελίτσκα, να περιμένετε λιγάκι να δείτε ε, πώς ε, θα εξελιχθούν αυτά τα συμβούλια. Εσείς είσαστε ιδιαίτερα ενεργός σε αυτό το τομέα, το έχω λάβει υπόψη μου και το θέμα έχει φτάσει σε επίπεδο πρώτου αντιπρόεδρου γιατί η Κομισιόν πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και αυτή για μένα είναι η πεμπτουσία των αρμοδιοτήτων μου και θα αποτύχω αν δεν τα καταφέρω καλά στο θέμα αυτό και με μεγάλη χαρά κύριε Τελίτσκα μετά εκ των υστέρων να μου ζητήσετε το λόγο, να με καταστήσετε υπόλογο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τίμερμανς για την παρέμβασή σας, ε, για την εισήγησή σας. Ε, προσβλέπουμε στις απαντήσεις και σας ξαναπερμένουμε με χαρά εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Good afternoon, dear colleagues, ladies and... Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Έχασα την ευκαιρία να ακούσω ε, τον Αντιπρόεδρο. Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να περιμένω μαζί με όλους τους άλλους ε, συνεπιβάτες μου δύο ώρες στη Φραγκούρτη γιατί δεν είχαμε διάδρομο για την πτήση μας και δεν μπόρεσα να είμαι εδώ στις αλλά είμαι σίγουρος ότι εγώ έχασα, δεν χάσατε εσείς. φτυχώς Δικό μου λοιπόν το πρόβλημα. Τώρα, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό, το επόμενο θέμα, που είναι ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τη ΜΜΕ. Στην Επιτροπή μας ε, είμαστε υπεύθυνοι για τις ΜΜΕ και γι' αυτό το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατατίθεται σε αυτή τη θητεία. Και η έκθεση κατατίθεται με βάση την, ε, ε, το σχέδιο της Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν κίνητρα αυτές ε, για να αναπτύξουν περτέρω την πράσινη ανάπτυξη. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Δεκέμβρη η Επιτροπή μας οργάνωσε ε, μια μεγάλη ακρόση για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Ε, πολύ σημαντική αυτή η ακρόση για τη δουλειά μας. Τώρα πια μετά την ακρόση γνωρίζουμε πολλά περισσότερα ως Επιτροπή και τη συζήτησή μας θα πρέπει να την έχουμε ολοκληρώσει σε μία ώρα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Ντεμπάκα είναι ο συγητής μας. Παρακαλώ συνάδελφε λοιπόν να μας ε, παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ο κ. Τίμερμαν θα μπορούσε να έχει βοηθήσει με αυτό το ζήτημα με το αεροδρόμιο που δεν είχατε χρονοθυρίδα, γιατί εκείνοι απέσυραν όλη την πρόταση για τι χρονοθυρίδε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά να σα παρουσιάσω σύστημα σήμερα την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την πρωτοβουλία για την πράσινη ανάπτυξη. Είχα πολλές συναντήσεις με πολλούς, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη για να προετοιμάσω αυτή την έκθεση και όλοι μου είπαν ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι περισσότερες, η πλειονότητα και έχουν πολλές ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να μεταβούν προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη οικονομία. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένοι, επομένως η βιωσιμότητα, η οικολογική βοηθά για τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Αρχές του Δεκεμβρίου είχαμε οργανώσει αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση και νομίζω ότι στην έκθεσή μου έχω συμπεριλάβει όλα τα θέματα που έθεσαν οι ε, ομιλητές εκείνη τη δημόσια ακρόαση καθώς επίσης και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι μετά οργανώσαμε επίσης και διάφορες συζητήσεις τρογγυλής τραπέζης με ομοσπονδίες ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και μιλήσαμε και με ε, επιχειρηματίες που μας εξήγησαν ποιες θα ήθελα να είναι οι κατευθύνσεις της πολιτικής μας καθώς επίσης και ποια μέτρα δεν θα έπρεπε να λάβουμε γιατί δεν λειτουργούν, δεν είναι αποτελεσματικά. Προσπάθησα λοιπόν εγώ να αποκρισταλώσω στην έκθεσή μου τις βασικές ιδέες που εξέφρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το ζήτημα για μένα δεν είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά για την πράσινη οικονομία, γιατί αν υπάρχουν άλλου είδους εμπόδια εξαιτία άλλων πτυχών της νομοθεσίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες Γι' αυτό στην έκθεση αναφέρομαι γενικά σε όλες τις δυσκολίες που αντιπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκινώ με τη δυναμική, με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεύτερον ε, είναι η χρηματοδότηση. Χρειάζεται επίσης ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και μια νομοθεσία κατάλληλη που να ευνοεί την καινοτομία. Είναι ξεκάθαρο ότι διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνούν ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε τι οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε στον τομέα της πράσινης οικονομία. Πρέπει να ε, φροντίσουμε να υπάρξει μείωση ε, των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται καθώς επίση και επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσή του, Θα αναφερθώ μόνο σε κάποια από τα κύρια ζητήματα. Ένα από τα κύρια θέματα που μου έθεξαν οι επιχειρηματίε είναι η έλλειψη η αδυναμία μάλλον ε, εξέβρεση χρηματοδότησης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει το ρίσκο και να αξιολογήσει και να καταλάβει, να αντιληφθεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορεί να προτείνει μια μικρομεσαία επιχειρήση. Πρέπει λοιπόν εδώ να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, τι περισσότερε φορέ οι τράπεζες, οι άλλοι πιστωτέ ε, επιδιώκουν, προσπαθούν με τα μοντέλα που, χρησιμοποιούν να μετρήσουν πώ μπορεί να μειωθεί το κόστος και δεν λαμβάνουν υπόψη του άλλου παράγοντε. Επίση, χρειάζεται ενίσχυση της διασυνοριακή συνεργασίας. Πολλέ φορέ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες Άρα πρέπει να βελτιώσουμε την διαφάνεια και να υπάρξει μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των ε, ομοσπονδιών ε, ενός κλάδου της βιομηχανίας οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και παρέχονται ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη τους. Το ζήτημα λοιπόν της πράσινης ανάπτυξης συνδέεται πολύ συχνά και με την ε, έρευνα και την κοινοτομία έναν τομέα στον οποίο είναι γνωστό ότι η Ευρώπη είναι μπροστά στον τομέα της βασικής έρευνας, αλλά όσον αφορά τη μεταφορά αυτής της επιστημονικής γνώσης στις πρακτικές εφαρμογές, εδώ υστερούμε. Και ίσως ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό δεν είναι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, γιατί είναι μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων που ε, αξιοποιούν δημόσια χρήματα για το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξής τους. Αντιθέτως, αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι ένα ε, επενδυτικό περιβάλλον και ένα σταθερό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο που να μην αλλάζει. Και αυτό θα οδηγήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά. Επίση, το ζήτημα τη ρύθμιση και της απορρίθμιση. Βάζουμε τρικλοποδία στον εαυτό μας. Ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα κράτη-μέλη ε, ε, ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομίζω δημιουργεί εμπόδια. Εάν χρειάζεται κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, αυτό πρέπει να είναι ευφυέ, πρέπει να είναι περιορισμένο στον τομέα των προμηθειών, για παράδειγμα των δημοσίων προμηθειών. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά επίσης χρειάζεται και μεγαλύτερη ε, ενημέρωση, έτσι ώστε να μην λαμβάνονται ε, ουσιαστικά από τους νομοθέτες, να, μην προκαταλαμβάνεται από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού από την ίδια την νομοθεσία και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών. Χρειάζεται επίσης βελτίωση του, των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των καταναλωτών, έτσι ώστε και οι ίδιοι καταναλωτές να προτιμούν τα προϊόντα που έχουν προκύψει από την πράσινη οικονομία. Θα έλεγα ότι έφυξα ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα της έκθεσής μου και βεβαίως θα συνεργαστώ και με τους συναδέλφους έτσι ώστε να καταλήξουν σε μια έκθεση η οποία θα είναι συνεκτική και ουσιαστική. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν σύντομο, συνεκτικό. Ε, Σα ευχαριστούμε πολύ. Τα αντιληφθήκαμε όλα και από πλευρά σε ΕΛΚ ο κύριο Κάριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια δήλωση από τον κύριο Ρούμπιχ, ο οποίο ε, δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα το απόγευμα. Επομένω ε, θα σα τη διαβάσω. Περιμένει και αυτός μια χρονοχωρηθυρίδα στη Βιέννη, φαντάζομαι. Κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, η ταπεινή μου ε, αναφορά τον όσων λέει ο κύριος Ρούμπιχ. Το ΕΛΚ ε, καλωσορίζει την προσέγγιση που ακολουθείται στην σχέδιο έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Ντεμπάκερ, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την υποστήριξη ε, ενός περιβάλλοντος που θα είναι βιώσιμο και... Ε, αποτελεσματικός προς τους πέρου, που θα δίνει όθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα αυξάνει τη δυνατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων που είναι απαραίτητα για τα διάφορα στάδια εξέλιξης μιας επιχείρησης. Πλέον των ε, φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό τη, θα πρέπει να υπάρχει και μια έγκαιρη εξέταση τη ε, ε, κείμενη νομοθεσία, χωρί να υπάρχει υπερβολική νομοθεσία και κανονισμοί από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει περιορισμό τη επαχθού νομοθεσία, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προσδώσει προστιθέμενη αξία. Ένα ελκυστικό ε, ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα είναι φιλικό προ τι επιχειρήσει και θα τι βοηθήσει όχι μόνο να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμε, αλλά και να αναπτυχθούν περαιτέρω και να έχουν μόχλευση στην ογετικό του ρόλο σε πράσινες τεχνολογίε, θα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επανεκβιομηχάνηση τη Ευρώπη. Αυτά λέει ο κύριο Ρούμπιχ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι συμφωνώ πλήρω με την άποψή του Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή έκθεση, ιδίω επειδή δίνει έμφαση στην μείωση της νομοθεσίας και το να μην υπάρχουν προσκόμματα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαρητήρια σας, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ σαφής παρατήρηση και τώρα ε, από ό,τι βλέπετε οι συντονιστές μας έχουν αναλάβει ε, ευθύνη για τις εκθέσεις. Ο κύριος Νίτσα τώρα, από πλευρά ε, σοσιαλιστών και δημοκρατών, ζητήσαμε από του συντονιστέ που δεν μπορούν να φύγουν ε, από τι Βρυξέλλε, γιατί δεν φοβούνται μήπω δεν έχει κατάλληλη χρονοθυρίδα. Μιλάω εξ ονόματο ε, του σκιώδη συζητητού για το θέμα. Έχει άλλο πρόβλημα, είναι σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση με τον Δανό Πρωθυπουργό, αλλά μπορούμε πάλι να πούμε ότι είναι θέμα χρονοθυρίδας. Καταρχάς, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το όσο ε, έχει κάνει στο θέμα αυτό και ε, θέτει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, κυρίως για την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότησή τους. Επειδή η χρηματοδότηση είναι σαφώς μια πολύ σημαντική πτυχή ε, για να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια υστέρηση σε αρκετούς τομείς που είχαν επισημάνει οι σκιώδεις εισηγητές κατά την αρχική συζήτηση που έγινε επί του ζητήματος. Από τις 3.000 ε, λέξεις που έχουμε στο σχέδιο κειμένου, περίπου 300 μόνο ασχολούνται με τη διαχείριση γνώσης, την έρευνα και την καινοτομία. Θέματα όπως για παράδειγμα αποτελεσματικότητας προς τους πόρους καλύπτονται απλώς σε κάποιες παραθέσεις και σε κάποιες αιτιολογικές σκέψεις και αναφέρονται μία φορά στο κείμενο στη βάση του κειμένου. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίε που θα μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Θα ήθελα να παρέμβω κι εγώ, γιατί είμαι εισηγητή για τη γνωμοδότηση για τι δυνατότητε πράσινη ανάπτυξη στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω τη σημασία του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να υποστηρίξω την αλλαγή προς μια ε, τοπική οικονομία σε όλους τους τομείς. Θα, αυτό θα συνάδει και με τους στόχους Ευρώπης 2020 για μια ε, ευφυή, βιώσιμη και ανάπτυξη που περιλαμβάνει τους πάντες θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους βασικούς μας στόχους και να ξεκινήσουμε πολιτικές οι οποίες θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε οικολογικές πολιτικές και πράσινη ανάπτυξη και θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Ελπίζω η γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Ρέτζη, στην οποία για την οποία θα γίνει συζήτηση την Πέμπτη, ε, θα ε, συμπεριληφθεί καταλήλως στην έκθεση της Επιτροπής Ήτρες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί ευχαριστούμε. Τώρα, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των ε, Ευρωπαϊκών Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών. Δεν ξέρω πού να είναι, στο αεροδρόμιο, στον Πρωθυπουργό. Επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Η ανακοίνωση επιτροπή μα λέει ότι το 3% των επιχειρήσεων καταβάλουν προσπάθειε για να προάγουν ε, την ε, σωστή χρήση των ε, πόρων. Μόνο οι 10 περίπου όμως, ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει σωστά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που προσφέρουμε και σε αυτό που εισπράττουμε. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο λειτουργούν τα μέτρα τα οποία διαθέτουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά πόσο είναι χρήσιμα τα μέτρα αυτά. Γνωρίζουμε ήδη ότι οι επιχειρηματίε καταβάλουν προσπάθεια για να επενδύσουν. Τώρα βιώνουμε κρίση και δεν νομίζω ότι κανεί το αμφισβητεί. Η δική μα λοιπόν δουλειά είναι να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στην αγορά και αυτό μπορεί να γίνει με χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όπω είπε και ο συγητή, με εγγυήσει, δάνεια, όλα αυτά δηλαδή τα οποία κατά κάποιον τρόπο στηρίζουν τις επιχειρήσεις που ήδη βρίσκονται στην αγορά, αλλά και όσοι θέλουν να μπουν στην αγορά. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να αλλάξουμε οπτική γωνία. Να ξεφύγουμε από μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στα χρηματοψηφικά και να γυρίσουμε σε μια πραγματική οικονομία. Δηλαδή να ε, δώσουμε νέα πνοή στον παραγωγικό ιστό. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο μέσω γραφειοκρατικής απλούστευσης, το ένα αν θέλετε, όχι μόνο, και το δεύτερο είναι ε, να καταστήσουμε ε, πιο αποτελεσματικές τις τοπικές διοικήσεις. Δηλαδή τα κονδύλια που παίρνουν να τα στοχεύουν, να τα χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη στόχευση και τα έμεσα κονδύλια να τα χρησιμοποιούν εξίσου αποτελεσματικά και τα έμεσα και τα άμεσα. Έτσι λοιπόν τα κονδύλια πρέπει να στοχεύουν σε εξειδικευμένες πράξεις με την έννοια ότι θα πρέπει να εντοπίζονται ποιοτικοί παράγοντες και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να φτάσει στην αριστεία δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε να ελέγχουμε και το αποτέλεσμα, γιατί αν λείπει αυτό το τελευταίο βήμα, νομίζω δεν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι σημαντικό. Άρα δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθούμε τι διαδραματίζεται και να επεμβαίνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε μια βιομηχανική παραγωγή η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις, ε, τις περιβαλλοντικές ανάγκες. Γιατί αν δεν το κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλικιώτης παρακαλώ εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχετε δίκιο τελικά οι συντονιστές αναγκαζόμαστε να λάβουμε τον ρόλο άλλων που απουσιάζουν. Ε, και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο για την καλή δουλειά που έκανε. Όμω ε, θα σημειώσω δύο-τρία ζητήματα. Ε, στο κείμενο δυστυχώ αγνοούνται ε, τα σκληρά μέτρα λειτουργία που επιβάλλονται, επηρεάζουν αντικά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και δεν αφήνουν περιθώρια ανάπτυξη καινοτομιών. γιατί έχουν αντιμετωπίσουν τεράστιου κινδύνου. Πρώτα-πρώτα είναι ο μεγάλο κίνδυνο απορρόφηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από μεγάλε πολυεθνικές. Ε, δεν γίνεται καμιά αναφορά ότι αναγκάζονται να πληρώνουν, να έχουν να δίνουν ψηλά επιτόκια, έχουν αδυναμία ανεξόφληση των χρεών του. και ε, τελικά ε, πάρα πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει καταλήγουν εν τέλει έρμενα των πιστωτών του με πολύ περιορισμένε δυνατότητες δράση. Και αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον στι χώρε του Νότου. Ε, και βεβαίως ε, θα, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να αναφέρουμε ότι η οικολογική καταστροφή οφείλεται εν πολύ στην ανεξέλεκτη δράση των μεγάλων εταιριών. Και γι' αυτό προκύπτει ανάγκη να στηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να λειτουργήσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Για μα, ένα πραγματικό σχέδιο στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα που έχουν να αντιμετωπίσουν και ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνε τι επιχειρήσει που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Στόχος θα πρέπει να είναι να δοθούν κίνητρα ανάπτυξη και απαραίτητα στηρίγματα που στερούνται σήμερα αρκετέ μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν διάφορες ε, ε, καινοτομίε και να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα προτεραιότητα μας λοιπόν θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση στις διαδικασίες πρόσβασης στη χρημαότηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να οθούν κίνητρα ανάπτυξη, να αυξηθούν τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για προγράμματα όπως ο Ορίζοντας 2020 και το Κόσμο Στο παρελθόν ασκήσαμε κριτική γιατί αντί να αυξάνονται μειώνονται αυτά τα κονδύλια και να δημιουργηθούν νέοι κανονισμοί για στήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των μεγάλων εταιριών. Εμεί ιδιαίτερα θέλουμε να δώσουμε ε, έμφαση στι πάρα πολύ μικρέ επιχειρήσει που αντιμετωπίζουν, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία που αντιμετωπίζουν και τι μεγαλύτερε δυσκολίε, ώστε όχι μόνο να προστατεύσουμε τις χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά α, ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Anybody from Greece? Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, κανείς? Δεν είμαι κανείς διαθέσιμος. Η κυρία Καηλή. Όχι, ο κύριος Κέλλη, συγγνώμη. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά ε, είναι ηρωνικό το γεγονό ότι συζητούμε δυνατότητε για πράσινη ανάπτυξη, μικρομεσαίες επιχειρήσει και δεν έχουμε εδώ πρασίνους να μα πούνε την άποψή του. Τέλο πάντων εμεί πρέπει να το προχωρήσουμε το ζήτημα και νομίζω ότι όπω ε, είπε και ο συνάδελφο Κάριν, πρόκειται για ένα πολύ λογικό και πρακτικό κείμενο και ο εισηγητή έχει καλύψει τα βασικά στοιχεία. Και κάπου πρέπει να υπενθυμίσουμε και στους εαυτούς μας ότι ε, η συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι συζητούμε για την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εάν δεν λειτουργούν καλά δεν θα έχουμε ούτε οικονομική ανάπτυξη, ούτε πράσινη ανάπτυξη, ούτε καμία ανάπτυξη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τις βοηθήσουμε. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να εξετάσουμε λίγο και τα όσα είπε ο κύριος Τίμερμαν, ο οποίο μα μίλησε προηγουμένω. κυρίω όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ανέφερε τι δυσκολίε που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει και το γεγονό ότι υπάρχει διάθεση πλέον να ασχοληθούμε με το ζήτημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν υπάρχει σχετικά εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν μπορούν να αναπτυχθούν και δεν μπορούν φυσικά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και το σχέδιο Juncker, εάν ξεκινήσει, που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, για την υπερβολική νομοθεσία και για το gold plating, την υπερβολική νομοθεσία και τους κανονισμούς σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι να ληφθεί υπόψη, διότι εάν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση σε εθνικό επίπεδο, ε, μπορεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορους τομείς ε, ε, της κυβέρνησης και να πρέπει να τους βρούμε αυτών θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται γενικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναζητήσουμε βέλτιστες πρακτικές. Δεν το κάνουμε αρκετά αυτό. Πολλά κράτη-μέλη ασχολούνται με τα δικά τους σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα καλύτερα και ελπίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ακριβώς δείχνει διάθεση να είναι λίγο πιο πρακτική και να σκεφτεί τι ακριβώς χρειάζεται, θα είναι σε καλή θέση να χρησιμοποιήσει αυτά τα βέλτιστα παραδείγματα και να τα δώσει ε, στους υπολείπους ώστε να μπορούμε να τα ρυθμίσουμε αυτά και σε επίπεδο κρατών μελών και γενικότερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί στη δέσμευση τη να έχουμε λιγότερη νομοθεσία και όχι περισσότερη νομοθεσία, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι βιώσιμη, ελκυστική και υποφελής για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και θα μπορούν να ασχοληθούν με την πράσινη ανάπτυξη, η οποία θα βοηθήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό σημείο κίνηση, ελπίζω να προχωρήσει και να έχει ωφέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλυτα δίκιο έχετε ότι δεν έχουμε μεταξύ μας κανένα από τους πρασίνους, αλλά Ευτυχώς, η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ντάντι, έχει μπροστά τη ε, πράσινη κάρτα, γιατί είναι αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής. Επιτροπή. Έχετε λοιπόν το λόγο, κυρία μου. Σημαντικό το ότι έχετε και πράσινη κάρτα. κανείς από τους πράσινους, αλλά έχει το πράσινη κάρτα μπροστά σας. Καταρχήν λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ε, νομίζω είναι ολοκληρωμένη η έκθεσή του και μου αρέσει το γεγονός ότι στην παράγραφο 22 αλλά και σε κάποια άλλα σημεία της έκθεσης υπογραμμίζεται την ανάγκη ε, να υπάρχει πιο επιχειρηματικό πνεύμα. Γιατί νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά στο σύνολο ε, δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά στο να προωτήσουμε και τους επιχειρηματίες και το επιχειρηματικό πνεύμα ανάμεσα στην νεολαία. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να ξεκινάμε ε, νωρίς με την εκπαίδευση ή να εξοικειώνονται με την επιχειρηματικότητα και τα συναφή θέματα. Πολύ θετικά λοιπόν όλα αυτά. Ε, θα ήθελα εκεί να αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι η ανάγκη να αναφερόμεθα σε μικροεπιχειρήσεις. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι μικροεπιχειρήσεις είναι μια πολύ σημαντική πηγή απασχόλησης. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές ε, μιλάμε γενικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι μικρές είναι τελείως διαφορετικές. Πρέπει να τους προσφέρουμε ε, τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Και αυτό απαιτεί και μια διαφορετική προσέγγιση για να προαχθεί η απασχόληση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια σχετική αναφορά στο σημείο υπαριθμών 4, αλλά θέλω το θέμα αυτό να προβληθεί περισσότερο ε, και πρέπει να προβληθεί περισσότερο στην έκθεση. Ήδη βέβαια είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ε, μια άμεση αναφορά στην παράγραφο υπαριθμών 4. Πρόεδρος, άλλος παρακαλώ επιθυμεί κάποιος άλλος το λόγο. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί την κυρία Τζοάννα Ντρέικ που είναι ε, Διευθύντρια ε, της Ανάπτυξης και των Μικρομεσαίων Επιχείρησεων της ε, Νέας Διεύθυνσης για την Ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τα μέλη και τους εισηγητές. Η Επιτροπή επιτιμεί να χαιρετήσει την ευρύτερη υποστήριξη που εκφράστηκε για την έκθεση. Και θέλω να σας πω ότι και εμείς συμμεριζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία να ληφθούν τα τα μέτρα και εποφελείς ε, κερδοφόρες ε, πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραμμα δράσης. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την ανταγωνιστικότητα. Οι μικρομεσαίες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι, κοστίζουν ε, πολύ ε, όμως οι μικρομεσαίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνες τους, αν προχωρήσουν μόνες τους δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε αυτό το πρόγραμμα, το πράσινο δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τι ευκαιρίες που υπάρχουν. Συγκεκριμένα υπάρχουν 34 δράσεις και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις ιδιαιτερότητες των μικρομεσαίων. Παραδείγματο χάρη, ε, ε, θέλουμε βελτίωση της επάρκειας πόρων μέσα στην ίδια την εταιρεία. Έχουμε την, ε, το επικείμενο κέντρο αριστείας για τη χρήση των πόρων. Εκεί θα προσφέρονται απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα ε, και τη σχέση κόστους ε, άμεσα αλλά και έμεσα μέσω συνεργασιών. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διευκόλυνση μεταφοράς τεχνολογίες ανάμεσα στις εταιρείες και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών προτύπων. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε και στο επιχειρηματικό σχέδιο για ε, διατομεακή προσέγγιση. Το πράσινο πρόγραμμα δράσης ε, μας επισημαίνει τους ε, μεσάζοντες ε, που έχουν αποδειχθεί χρήσιμη στην πράξη όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά και συνεργατικοί σχηματισμοί που διευκολύνουν τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική ανάληψη εργασιών το πρόγραμμα δράσης βασίζεται στο πώς οι στρατηγικοί συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να αποτελούν εργαλείο για να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, πάντα για ΜΜΕ και κυρίως ε, τις ανησυχίες που έχουν οι ΜΜΕ. Εμείς στηρίζουμε και συμφωνούμε με την έκθεση ότι οι μικρομεσαίες έχουν συγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές ανάγκες που αποτούν και συγκεκριμένες λύσεις ας πούμε με τη μορφή ενός ευρύτερου φάσματος χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ας πούμε η περίοδος από το 14 στο 20 εκεί η πράσινη ανάπτυξη αφορά τη χρηματοδότηση για εργαλεία τα οποία θα αντιμετωπίζουν την περιορισμένη πρόσβαση σε εμπορική χρηματοδότηση για επενδύσεις που εξοικονομούν ενέργεια. Επίσης ε, και άλλες διευκολύνσεις που χρηματοδοτούν προγράμματα της ε, βιοπικιλότητας μεταξύ άλλων οι μικρομεσαίες μπορούν να επωφεληθούν και από αυτό που λέμε ε, χρηματοψηφικό εργαλείο COSME. Είναι οι ε, διευκολύνσεις για ανάληψη πιστώσεων μεταξύ άλλων. Εμείς λοιπόν έχουμε ενισχύσει ε, και το, χρηματοψηφικό, το μετοχικό χρηματοψηφικό εργαλείο. Μάλιστα έχει υπάρξει και ένα θέμα που αφορά στην ενημέρωση. Έχουμε συστήσει μια πύλη, χρηματοψητική πύλη, που διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρόσφατα έχει συστήθει αυτή η πύλη και εκεί συγκεντρώνονται όλες οι πηγές ε, πληροφόρησης για τη χρηματοδότηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και έτσι λοιπόν όποιοι ΜΜΕ ή όλες έχουν πρόσβαση σε αυτή την πύλη και μου είπαν μάλιστα σήμερα ότι σε αυτή την πύλη είχαμε ε, και έχουμε περίπου 100.000 χτυπήματα το μήνα και το 60 κάτι είναι τακτικοί χρήστες. Πολύ καλό αυτό το νέο και θέλουμε να συμπεριλάβουμε και πηγές χρηματοδότησης και από τα αντιερθρωτικά ταμεία. Πάντα βέβαια για τις ΜΜΕ. Όλες αυτές οι χρηματοψηφιακές δυνατότητες περιλαμβάνουν ε, και προγράμματα για καθαρή τεχνολογία. Ενδεικτικά το λέω. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια εξαρτία ενημέρωση για τα κρατημέλη και τους άμεσα εμπλεκόμενους και εκπαίδευση για συμβούλους έτσι ώστε να ενισχυθεί η δραστηριότητα των χρηματοψηφιακών συμβούλων που είναι η καλύτερη βοήθεια επιτόπου. Τέλος, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το 1 τέταρτο των κονδυλίων του θα το δώσει για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές και οι μεσαίες κεφαλοποίησης, να αναπτυχθούν. Εξάλλου, το πρόγραμμα ε, θα στηρίξει και προγράμματα ε, φιλικά προς το περιβάλλον. Όσον αφορά τη νομοθεσία, χάρηκα που άκουσα την ομιλία του κυρίου Τίμερμανς, βεβαίως και πρέπει να ε, περιορίσουμε τη γραφειοκρατία ε, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Και μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος ε, Τίμερμανς, δηλαδή μίλησε για κάποια πολυπλοκότητα του συστήματος. Προφανώς το θέμα των ΜΜΕ πρέπει να είναι πιο ορατό, ένα αναπόσπαστο στοιχείο των διαδικασιών ανάλυσης επιπτώσεων. Αυτά ε, σημαίνουν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως θεωρώ ότι πρέπει να τα προβάλλουμε περισσότερο τα θέματα. Και υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία προχωράνε στις βέλτιστες πρακτικές. Τελειώνοντας, η Επιτροπή χαιρετίζει την ευρύτερη υποστήριξη αλλά και τη φιλοδοξία να υπάρχουν κατάλληλες ενέργειες για να στηριχτούν κερδοφόρες πρωτοβουλίες. Εμείς ε, προσβλέπουμε στην ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην εφαρμογή ε, του πράσινου προγράμματος δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την παρουσίαση για το σχέδια διαδράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Ανάπτυξη. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, το... να δώσω μάλλον το λόγο στον συνάδελφο Ντεμπάκερ για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Κύριε Ντεμπάκερ, ναι, θα είμαι σύντομος γιατί από φαίνεται έχουν ικανοποιηθεί όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για όλες τις ιδέες και τις ε, παρατηρήσεις που έκαναν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε τι τροπολογίε που υποβάλλονται όχι μόνο σε αυτή την Επιτροπή αλλά και στις υπόλοιπες μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξετάσω προσεκτικά τα σχόλια που μου κάνετε. Δεν θα δυσκολευτούμε νομίζω να βρούμε συμβιβαστική λύση και να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα καλύπτει και τις δικές σας παρατηρήσεις. Τελικά να καταλήξουμε σε μια έκθεση προς την Επιτροπή η οποία θα είναι ξεκάθαρη έτσι ώστε να ξεκινήσει και η υλοποίηση. Κάτι που πρέπει να γίνει επίση και στο επίπεδο των κρατών μελών. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφα για αυτή την παρουσίαση και να σας υπενθυμίσω ότι, ότι 26 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 12 το μεσημέρι, προφανώς, 26 Φεβρουαρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή, αυτή τη βδομάδα. Με αυτά λοιπόν κλείσαμε και το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Το επόμενο 13 λεπτά μας πήρε. Το επόμενο λοιπόν σημείο είναι η συνάντηση των συντονιστών. Μάλλον έχετε 13 λεπτά στη διάθεσή σας για να φύγετε από την αίθουσα εάν δεν έχετε δικαίωμα να παρευρεθείτε στη συνάντηση των συντονιστών. Άρα δεν βιάζεται κανένας. Σιγά σιγά.